Καλημέρα σας, καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. Ας ε, καλωσορίσουμε τον Υπουργό Στερικών της Ισπανίας, τον Αλφρέντο Πέρες Ρουμπαλκάμπα. Καταρχάς θα κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Στα ισπανικά. Μετά την χθεσινή αναθεώρηση που έγινε στο Συμβούλιο, για το σχέδιο απόφασης όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρόκειται για τη συμφωνία TFTP, Σύστημα Οικονομικού Εντοπισμού Τρομοκρατών, σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Στο σημείο μάλλον 10 της ημερήσιας διάταξης θα επικεντρωθούμε στο ζήτημα αυτό. Στο σημείο 11 τώρα της ημερήσιας διάταξης, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας, Το σημείο αυτό θα το συζητήσουμε μετά το σημείο 8. Το σημείο 8 που έχει ως θέμα τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης. Αυτό προβλέπεται για τις 10 αύριο το πρωί. Τώρα το σημείο 12 στη μερίσια διάταξη Το σημείο αυτό έχει να κάνει με την οδηγία για την νήση μεταχείριση των προσώπων, για την ε, κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης και έχει αναβληθεί για τις 4 Φεβρουαρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τις αλλαγές αυτές στην μερίσια διάταξη μπορούμε να την εγκρίνουμε. Όσοι ενδιαφέρει τώρα για τη συζήτηση που θα γίνει για τα σκάνερ σώματος, τους ανιχνευτές. Η Επιτροπή Μεταφορών θα συζητήσει το ζήτημα αυτό αύριο το απόγευμα. Όσοι λοιπόν από την ε, Επιτροπή μας ενδιαφέρεστε μπορείτε σαφώς να πάτε στη συζήτηση αυτή που θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή Μεταφορών είναι η αρμόδια για τη συζήτηση του ζητήματος του οποίου αναφερθήκατε, έτσι δεν είναι, Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν έχει δοθεί οριστική εντολή αυτή τη στιγμή. Δεν έχει δοθεί επίσημα και αποκλειστικά η συζήτηση για τους ανιχνευτές σώματος στην ε, Επιτροπή Μεταφορών. αλλά προβλέπεται να συζητηθεί το ζήτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη την αυριανή της Επιτροπής Μεταφορών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν μου το επιτρέπετε, να σας ευχαριστήσω μάλλον και να σας ζητήσω να υποβάλλετε γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Μεταφορών. Πρόεδρος, ναι, ναι, το σημειώνουμε αυτό το έτοιμά σα Πάντως, ε, η Επιτροπή Μεταφορών μας ενημέρωσε ότι όσοι επιθυμείτε να πάτε στην ευρενή τη συζήτηση είστε ευπρόσδεκτοι αύριο το απόγευμα. Τώρα, όσον αφορά περαιτέρω τις ανακοινώσει του Προέδρου, θα ήθελα να υποστηρίξω την απόφαση των ε, συντονιστών να διορίσουμε τον κύριο Βιν Βαντεκάμπ ω εισηγητή για την ε, συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της ε, Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Λίχτενστάιν. Συμφωνία που έχει να κάνει με τους επιπλέον κανόνες σε σχέση με το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ε, η κυρία Λάτφορντ που είναι η συγγήτρια για το θέμα εκείνο που έχει να κάνει με την μετάφραση και τη διερμηνία και η κυρία Χέτθ και η κυρία Αντζελίνη επιβεβαιώνονται. Η κυρία Χέτθ για την ε, εμπορία ανθρώπων και η κυρία Αντζελίνη για την παιδική πορνογραφία. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κάσμαν, πρώην εισηγητής για τον κώδικα συνόρων Σέγγεν, έχει εξετάσει ένα σχέδιο πρότασης ε, του Συμβουλίου όσον αφορά την επιτήρηση των συνόρων και όπως αυτή συντονίζεται από τη Frontex. Πρόκειται για ένα μέτρο επιτροπολογίας και συζητήθηκε στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Καθότι λοιπόν το Συμβούλιο ενέκρινε την επίσημη θέση του χθες, το Κοινοβούλιο έχει πλέον δύο μήνες για να προτιμάσει τη θέση του. Ο κύριος Κάσμαν λοιπόν προτείνει να υποβληθούν ορισμένες ερωτήσεις προς την νομική υπηρεσία προκειμένου να διευκρινιστεί αν όντως η επιτροπολογία είναι η ακολουθητέα η καλύτερη δυνατή διαδικασία για το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις θα προωθήσουμε τα ερωτήματα αυτά, το ζήτημα αυτό προς την νομική υπηρεσία. Κύριε Κάσμαν, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, δεν θέλω να σας καθυστερήσω ετοίμασα ένα φάκελο για, τα, για τους βουλευτές με δύο ερωτήσεις προς την νομική υπηρεσία. Σήμερα ήρθα σε επαφή με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν για να συζητήσουμε τις προτάσεις τους και νομίζω ότι θα πρέπει να δράσουμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε μια προθεσμία δύο μηνών, μέσα στην οποία το Κοινοβούλιο πρέπει να απαντήσει. Ευχαριστώ. Το σημειώνουμε, κύριε Κάσμαν. Και τώρα σας συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο, που είναι η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς του Υπουργού Εσωτερικών της Ισπανικής Κυβέρνησης. Τον κύριο Αρφρέντο Περές ε, Ρουμπαλκάβα. Θα ήθελα ο Υπουργός να χρησιμοποιήσει 15 λεπτά για να κάνει την παρουσίασή του. Εν συνεχεία θα ακούσουμε ερωτήσεις και θα απαντήσει ο υπουργό. Δύο λεπτά θα δοθεί στην κάθε ερώτηση και δύο λεπτά στην κάθε απάντηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία τώρα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να αυτοπεριοριστείτε, να είστε λακωνικοί, ούτως ώστε να έχουμε όλοι χρόνο να μιλήσουμε. Ο κύριος υπουργό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές. Για πρώτη φορά έρχομαι στην Επιτροπή σας και στο, Κοινοβούλιο για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Καθότι εμείς είμαστε... Έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Τζάι και θα την έχουμε για το πρώτο εξάμεινο του 2010. Τέταρτη φορά έχουμε την Προεδρία από πλευράς Ισπανίας και γνωρίζουμε ότι τα διακυβεύματα είναι πολύ σημαντικά και έχουμε ετοιμάσει το πρόγραμμα με τις δύο χώρες που θα ακολουθήσουν στην Προεδρία, την το Βέλγιο και την Ουγγαρία. Ετοιμάσαμε λοιπόν αυτό το πρώτο πρόγραμμα με τρόπο σοβαρό και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να υλοποιήσουμε τις, ε, τους στόχους που έχουμε θέσει για τη δική μας Προεδρία και τις δύο επερχόμενες. Είναι μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Μια νέα επιτροπή θα διοριστεί και ξέρετε ότι οι δύο τομείς ε, εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικοί Επίσης, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα μας καθοδηγήσει στην Ισπανική αυτή Προεδρία σε ό,τι αφορά την πολιτική εσωτερικών υποθέσεων. Μία από τις πρώτες συνέπειες της θέσης ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας είναι η πιο έντονη παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεσμικό πλαίσιο. Έτσι το θέλησαν οι Ευρωπαίοι. Όλα τα θεσμικά όργανα το θέλησαν επίσης και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε τόσο ώστε να, να συνδέσουμε πιο άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτε με τα θεσμικά τους όργανα. Και σε αυτή την περίπτωση μιλώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο στόχος μας λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να πω τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι ευχή κάνω, τι επιθυμίες έχω σε ό,τι αφορά τους έξι επόμενους μήνες. Θα ήθελα να συνεργαστούμε τους έξι μήνες και να υπάρξει συνένεση για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναδείξει τη συναπόφαση σε μια τακτική συνηθισμένη διαδικασία στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και είναι η λογική συνέπεια της εξάλληψης του τρίτου πυλώνα. Μία από τις συνέπειες είναι ότι όλες οι αποφάσεις του χώρου εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης περνάνε στον τομέα μας, στην ε, τακτική διαδικασία. Είμαστε ικανοποιημένοι που η συνθήκη της Λισαβόνας εντάσσει και την ε, Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η μεγάλη κατάκτηση του διεθνούς δικαίου πολεμικά εντάσσεται πλέον και στη δική μας νομοθεσία, δημιουργώντας και υπογραμμίζοντας τις αξίες που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα στοιχεία μέσα στα οποία, τα οποία δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Θα θέλαμε λοιπόν το πρόγραμμά μας να λάβει υπόψη όλα αυτά τα νέα στοιχεία. Και η βασική στόχοι είναι η ασφάλεια των πολιτών να γίνει να προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει ε, προστιθέμενη αξία για αυτήν. Θα θέλαμε λοιπόν η να εστιάσουμε στην ασφάλεια των πολιτών και όλες οι πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσουμε σήμερα το απόγευμα έχουν σαν στόχο να αισθανθούν όλο και πιο σίγουροι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ούτω ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και τις ελευθερίες τους. Η ασφάλεια στο βωμό της ελευθερίας και η ασφάλεια σέβεται όλες τις αρχές της ελευθερίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο πολύ σωστό πλαίσιο που έθεσε και η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα αναφερθώ στις πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουμε τους επόμενους έξι μήνες. Ε, θα τις διαρρέσω σε τρεις άξονες. Καταρχάς αυτοί οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα με υποχρεωτικό τρόπο. Επίσης θα παρουσιάσω τις ισπανικές πρωτοβουλίες και ο τρίτος τομέας, το τρίτο πακέτο είναι ένα σύνολο πρωτοβουλειών με πιο άμεσο χαρακτήρα που στόχο έχουν να ενδυναμωθεί η αστυνομική συνεργασία στον ευρωπαϊκό χώρο. Επομένως, καταρχήν θα μιλήσω για τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναπτύξουμε τους έξι επόμενους μήνες και που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που τέθηκε σε ισχύ, και τώρα απόκειται στην Κομισιόν να προτείνει στο Συμβούλιο το σχέδιο δράσης που απορρέει από το πρόγραμμα τη Στοκόλμης. Αυτό θα αποτελέσει δουλειά του Συμβουλίου τους επόμενους έξι μήνε και θα θέλαμε να υιοθετηθεί τους έξι πρώτου μήνε του 2010, μέσα, κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο εξάμεινο λοιπόν. Προτείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δουλέψουμε εκ του σύνεγγυ, ούτως ώστε αυτό το σχέδιο ε, δράσης να αντιπροσωπεύει και τους στόχους, τις ανησυχίες και τα μελήματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τους έξι πρώτους μήνες επίσης του 2010 θα κάνουμε μια αποτίμηση του α, συμφώνου για το άσυλο και την μετανάστευση που υιοθετήσαμε το 2008. Δεν πρόκειται για αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ο συνάδελφος εν συνεχεία θα υπησέλθει σε λεπτομέρειες. Εν συνεχεία η Ισπανική Προεδρία θα συνεχίσει την εξέταση κάποιων φακέλων, κυρίως αυτών που συνδέονται με την εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών, του ΣΥΣ και του ΒΙΣΑ. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό κοινό σύστημα ασύλου. Είμαστε ικανοποιημένοι διότι καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν, τόσο ώστε να δημιουργήσουμε το γραφείο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για το άσυλο. Οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και επομένως στου έξι πρώτους μήνες του 2010 θα ιδρύσουμε στη Μάλτα όπως αποφάσισε το Συμβούλιο αυτό το γραφείο για το άσυλο. Εν συνεχεία έχουμε το, πρόγραμμα επανεγκατάστασης και ελπίζουμε τους, το πρώτο εξάμεινο του 2010 να έχουμε ένα πρόγραμμα ειδικό επανεγκατάστασης που θα είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και εξελιγμένο. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στους υπόλοιπους φακέλους ε, οδηγιών και κανονισμών που έχουν μια επίπτωση στο Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ορίμανση εντό αγωγικών αυτών των φακέλων και ίσω δεν θα μπορέσουμε το πρώτο εξάμεινο του 2010 να κλείσουμε όλου του φακέλου. Θα θέλαμε όμω να προχωρήσουμε στι συζητήσει ούτω ώστε οι Βέλγοι συνάδελφοι εν συνεχεία να ολοκληρώσουν αυτό το πακέτο μέτρων που θα μα επιτρέψει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και να έχουμε τον επόμενο χρόνο ένα κοινό σύστημα ασύλου. Εν συνεχεία, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου ε, θα προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες του συς και του ΒΙΣ. Θα ξέρετε ότι το ΣΥΣ2 ε, προσκρούει σε κάποια προσκόμματα αυτή τη στιγμή. Ε, αυτή τη στιγμή κάναμε μία αξιολόγηση της λειτουργίας του, κάτι που είχαμε συμφωνήσει ούτως ή άλλως πριν από λίγους μήνες και με βάση αυτό τον απολογισμό θα έχουμε τώρα δύο μήνες στη διάθεσή μας για να δούμε εάν θα συνεχίσουμε τι δραστηριότητε, στα πλαίσια του ΣΥΣ2 ή αν θα εμβαθύνουμε το ΣΥΣ. Θα ήθελα να ρυθμίσουμε το, πρόβλημα του ΣΥΣ2 και θα ήθελα να σα πω ότι θα σα ενημερώσουμε, θα σα κρατούμε ενήμερου εσά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα τα στοιχεία που θα αλλάξουν, για όλη την πρόοδο που θα σημειωθεί. Ούτω ή άλλω είναι μια πρωτοβουλία τη Κομισιόν σε ό,τι αφορά αυτό το σύστημα ενημέρωση. Για το σύστημα θεωρήσεων τώρα, το ΔΙΣ, είναι ένα πολύ σημαντικό σύστημα που ο σκοπό έχει να, γίνουν πιο διαφανείς οι πολιτικές μας για τις θεωρήσεις. Αυτό το σύστημα, το ΒΙΣ, θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του 2010. Αντιμετωπίζουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες ε, στα πλαίσια, όπως σας είπα, του ΣΥΣ2, αλλά αυτές είναι άσχετες με το σύστημα ΒΙΣΕ. Ε, πιστεύουμε ότι το σύστημα VIS τεθεί σε ισχύ εμπρόθεσμα. Ε, δεσμεύομαι ενώπιον τη Επιτροπή σα να σα ενημερώνω για όλε τι προόδου, για όλε τι εξελίξει για το σύστημα VIS. Επίση, θα ήθελα σε ό,τι αφορά αυτό το πρώτο πακέτο ας πούμε, θεμάτου, ε, να σας πω ότι η συνθήκη μας υποχρεώνει να δημιουργήσουμε μια επιτροπή εσωτερικής ασφάλειας, ούτως ώστε να ενθαρρύνουμε την εσωτερική συνεργασία Κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας θα δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα και θα θέλαμε αυτή η Επιτροπή είναι ένα σημείο κλειδί, ένα όργανο κλειδί, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα, δηλαδή ότι όλα τα, όλοι οι φορείς που προωθούν την ε, ασφάλεια ε, συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα θα περάσω στις πρωτοβουλίες που ονόμασα στην αρχή της παρουσίασής μου το δεύτερο πακέτο, ας πούμε, η δεύτερη δέσμη πρωτοβουλειών. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που η Ισπανική ε, Προεδρία θεωρεί ότι είναι στρατηγική σημασία ε, και πέρα από τη δική μα Προεδρία, πέρα από το εξάμεινο τη προεδρία μα, Αυτού του έξι μήνες θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα, ένα έγγραφο που θα συνδέεται με τη στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια. Μια στρατηγική η οποία αναφέρεται ήδη στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Σε τι συνίσταται αυτή η στρατηγική τώρα. Τι θα θέλαμε να συμπεριλαμβάνει αυτό το έγγραφο. Θα θέλαμε να είναι ένα λακωνικό, ένα συνοπτικό έγγραφο, το οποίο με εύληπτο τρόπο εξηγεί στους Ευρωπαίους πολίτες ποια, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιες είναι οι απειλές, στις οποίες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύμφωνες. Σε μια δεύτερη φάση θα θέλαμε να τους εξηγήσουμε τι πρόοδο έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια σε θεσμικό επίπεδο, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι απειλέ και του κινδύνου. Εδώ έχω υπόψη μου τη Europol, τη Eurojust, τη Frontex και προφανώ ε, και τη θέση σε ισχύ α, ε, τις του συντονιστή για, τον, για την τρομοκρατία. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μοντέλο της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ε, ξεκινώντας από την ε, πρόθεση όλων των αξιών που στηρίζουν, όπου εδράζεται αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, οι ατομικές ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών. Τέταρτον, πιστεύουμε ότι αυτή η στρατηγική, σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να βασίζεται στις 10 θεμελιώδεις ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, πάνω στις οποίες εργάζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους και τις απειλές ε, που και εμείς αλλά και οι άλλες χώρες. Απειλές που εναντίον μας αλλά και άλλων χωρών. Θα θέλαμε λοιπόν να υιοθετήσουμε, να σας μιλήσουμε για αυτό το θεσμικό μηχανισμό που έχει ήδη συσταθεί, αλλά θέλουμε να τον βελτιώσουμε. Θα θέλαμε να εξηγήσουμε στους πολίτες την στρατηγική μας για την ασφάλεια και θα θέλαμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι ανησυχίες τους και τα προβλήματά τους αντικατοπτρίζονται στον τρόπο λειτουργία των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Με αυτές τις ανησυχίες ε, για τα θέματα ασφάλειας θα θέλαμε να δώσουμε και μία όθηση στις διατλαντικές σχέσεις. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι σχέσεις. Πρόσφατα υπήρξε ένα παράδειγμα των κοινών απειλών που αντιμετωπίζουμε ε, το ζήσαμε αυτό, την απόπειρα, την πρόσφατη, την πρόσφατη απειλή έχω υπόψη μου, αυτήν εννοώ, και ξέρω πολύ καλά ότι ο, ίσως, ο Ισλαμικός παραμένει μια σημαντική απειλή και ο στόχος του είναι να πλήξει την ε, εμπορική μας αεροπορία. Θα ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου που έλαβε χώρα στον, στο Τολέδο μαζί με την Αμερικανή ε, Υπουργό κυρία Ναπολιτάνο, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας που στόχο έχει να ασχοληθεί με αυτά τα πολύ συγκεκριμένα θέματα που είναι και πολύ ανησυχητικά για τους πολίτες μας και την κοινή γνώμη. Πώς θα βελτιώσουμε δηλαδή την ασφάλεια στα αεροδρόμια και δεν εννοώ μόνο τα αεροδρόμια, αλλά εννοώ και στα, μέσα στα αεροπλάνα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα ελέγχου των εκρηκτικών και το σύστημα ανταλλαγής των πληροφοριών, τις δυνατότητε έρευνας, τις τεχνολογικές δυνατότητες για να προωθήσουμε την έρευνα και τα σχέδια συνεργασίας με τις τρίτες χώρες που συχνά ε, είναι τα ορμητήρια ε, των τρομοκρατών. Θα θέλαμε αυτός ο τομέας του, της Ισλαμικής τρομοκρατίας να μην ε, είναι ο μονός τομέας στον οποίο θα στηρίζονται οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θέλαμε να έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο βελτιωμένες σχέσεις για να καταπολεμήσουμε την ε, διασυνοριακή εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και θα διενεργήσουμε υπουργικές συνεδριάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και δικαιοσύνη από πλευρά Ευρώπη και Αμερική που θα γίνει τον Απρίλιο και εκεί θα προτείνουμε ε, τον εξή στόχο, να ενδυναμώσουμε αυτόν τον διατλαντικό χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνη. Τέλος, θα ήθελα να περάσω σε ένα σύνολο θεμάτων ε, για να καταλήξω που όπως είχα πει στην αρχή ανήκε στο τρίτο άξονα θεμάτων που θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και που θα μπορούσα να κυκλοφορήσω ε, πρωτοβολίες για να βελτιώσουμε την επιχειρησιακή μας συνεργασία. Δηλαδή, ε, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ε, μηχανισμών και δυνάμεων ασφάλειας και φορέων ασφάλειας. Έχουμε την πρόθεση να δούμε τι είδους συνεργασία θα μπορούσαμε να έχουμε, ώστε όλες οι αστυνομικές δυνάμεις να συνεργάζονται. Θα πρέπει η αστυνομία να έχει εμπιστοσύνη και επομένως θα πρέπει να εμβαθύνουμε στις μεθόδους ε, ενημέρωσης μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κοινέ δυνάμεις συνεργασίας όπως υπάρχουν στην απόφαση Πλουμ και να διευκολύνουμε τους ε, μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αστυνομιών ή αστυνομικών δυνάμεων και θα υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα έρασμος για τις αστυνομίες που σκοπό έχει να ε, εντάξει τις εμπειρίες στα προγράμματα κατάρτισης, εμπειρίες που είναι θαυμάσιες στον τομέα της ε, παιδείας ε, με τους φοιτητές που ανταλλάσσονται από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο με αυτό, αυτό θα το εφαρμόσουμε τώρα σε αστυνομικό επίπεδο για να ενδυναμώσουμε την αστυνομική συνεργασία. Ε, αυτή η ενδυνάμωση θα λάβει χώρα σε διάφορους τομείς της καθημερινής μας δράσης που συνδέεται με την τρομοκρατία και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδη στοιχεία, ε, θεμελιώδης ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αναφέρθηκα στι ΗΠΑ. θα θέλω να σα πω ότι κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα θα παρακολουθήσουμε αυστηρά τι στρατηγικέ μα και τα σχέδια δράση μα. Αυτά που έχουμε για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Ακριβώ γι' αυτό θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο των εκρηκτικών, ούτω ώστε να έχουμε ένα σύστημα ε, προειδοποίηση μεταξύ των χωρών μα και επίση θα δημιουργήσουμε και ένα σύστημα που στόχο έχει να δημιουργηθεί ε, μια ίχνη λασιμότητα σε ό,τι αφορά το ενδοκινοτικό εμπόριο εκρηκτικών υλών. Και επίσης θα δημιουργήσουμε ομάδες με τρίτες χώρες που θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθειά μας και θα δημιουργήσουμε επίσης μηχανισμούς συντονισμούς ε, στα πλαίσια των πυρήνων συντονισμού που έχουμε σε εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα προβούμε και σε μία ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στο τομέα της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική, υπάρχει ένα πρόγραμμα σε κάθε μία από τις χώρες μας που σκοπό έχει να προωθήσει διάφορα μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ότι μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε μέσα στους ΔΕΣ. Ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, είναι σαφές ότι όλα τα δεδομένα, ότι όλες οι αναλύσεις της Europol ε, δείχνουν ότι μια άλλη μεγάλη απειλή είναι το οργανωμένο έγκλημα και θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε την ε, την, εγκληματικότητα δηλαδή στον κυβερνοχώρο, στο διαδικτύο. Και επίσης και το ξέπλυμα του χρήματος. Θα δούμε πώς ε, θα διαχειριστούμε τα, τις προσόδους ε, από παράνομες δραστηριότητες. Θα δουλέψουμε με πράκτορες ε, σύνδεσης που δραστηριοποιούνται στη Σενεγάλη, στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Λατινική Αμερική για να δούμε πώ θα προωθήσουμε τι στρατηγικέ μα. Θα στηρίξουμε την Europol επίση και βεβαίω θα ασχοληθούμε ξανά με το οργανωμένο έγκλημα για να το καταπολεμήσουμε με τη δημιουργία ενός δικτύου που προέκυψε από δύο πρωτοβουλίες. Μία που συνδέεται με τις γυναίκες και μία άλλη που συνδέεται με τις γυναίκες, με, με Νομίζω ότι πρέπει να τα σκεφτούμε πιο σοβαρά αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε τη γενική μας προσέγγιση. Αυτό συνδέεται με το σύμφωνο που ανέφερα προηγουμένως, ότι θα θέλαμε να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας με τις χώρες που αποτελούν ορμητήριο τρομοκρατών, ε, Θα πρέπει να συνδέσουμε την ε, μετανάστευση με μια πολιτική η οποία θα μας επιτρέπει να προωθήσουμε την νόμιμη μετανάστευση και να καταπολεμήσουμε τη λαθομετανάστευση. Θα ενδυναμώσουμε τη Frontex. Πιστεύουμε ότι πρέπει να τη στηρίξουμε περισσότερο από πλευράς, ε, να στηριχθεί περισσότερο από πλευρά κομισιών πιο συγκεκριμένα, ούτω ώστε να ευοδοθούν αυτοί οι στόχοι. Επίσης θα θέλαμε να ασχοληθούμε και με την ε, καταπολέμηση της πλαστογράφησης των ε, ταξιδιωτικών εγγράφων και των άλλων επισήμων εγγράφων. Θα καταπολεμήσουμε βεβαίως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Έχουμε ήδη σημειώσει θετικά βήματα στην ε, Λισαβόνα, στην Άκρα, στη Σενεγάλη και θα θέλαμε να δυναμώσουμε και να παγιώσουμε αυτές τις πρόοδους θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το νέο δρόμο της κοκαίνης ε, που περνάει μέσα από τη Δυτική Αφρική. Τέλος, θα θέλαμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε δύο ή μάλλον τρία θέματα που κατά την άποψή μας αξίζουν ε, περαιτέρω προβληματισμού στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου. Πρόκειται για τη βία την ε, οικιακή, τη βία μεταξύ των φίλων, αν θέλετε, από τους άντρες προς τις γυναίκες. Ε, πρέπει να κάνουμε μια, μια κοινή σκέψη. Εδώ συνδέεται αυτό το θέμα με την πολιτική και αστική προστασία. Ε, επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με την πρόληψη των πυρκαγιών και τις πρακτικές για να βελτιώσουμε την ασφάλεια στους αυτοκινητοδρόμους. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές του προγραμματός μας, το οποίο είναι φιλόδοξο, αλλά πιστεύω ότι είναι και ρεαλιστικό παράλληλα. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπα στην αρχή, ότι θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και όλος ιδιαίτερος με το κοινοβούλιο σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές για την προσοχή σας. Gracias, ministro. Τώρα θα ξεκινήσουμε με το γύρο των αεροτοαποκρίσεων. Έχω ήδη ένα μακρύτατο κατάλογο μελών της Επιτροπής μας που ζήτησαν το λόγο. Ε, ο μέγιστος λόγος ε, για κάθε ερώτηση και κάθε απάντηση θα είναι δύο λεφτά. Το υπενθυμίζω, έτσι. Ε, παρακαλώ όλοι να είσαστε λακωνικοί, ούτω ώστε να μπορέσουν να πάρουν το λόγο ώστε να τον περισσότεροι βουλευτές το χρόνο που έχουμε. Ο πρώτος και καλύτερος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τις καλύτερες μου ευχές στην ε, Ισπανική Προεδρία για το νέο έργο της. Και θα ήθελα να έχω μια διευκρίνηση κύριε Υπουργέ σε σχέση με τις Ισπανικές Προεδρίες, με τις προτεραιότητές σας. Έχετε πει ότι είσαστε εναντίον της βίας κατά των γυναικών και υπέρ της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά υπάρχουν και άλλα θύματα στην κοινωνία μας, είναι τα θύματα της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω την δέσμευση του Επιτρόπου Μπαρό να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Χάρτα για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν είναι της αρμοδιότητάς σας ε, απολύτως, αλλά έχουμε τρεις καυτές πατάτες ούτως υπήν. Θέλουμε να προστατεύσουμε τις ε, δημόσιες ελευθερίες. Έχουμε το SWIFT, έχουμε τα PNR για τις αεροπορικές συγκοινωνίες και έχουμε και τους body scanners, τους αρωτές σώματος. Εγώ συμφωνώ με το να υπάρχουν κοινέ ομάδες για αστυνομική συνεργασία αλλά είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί για ένα τέτοιο θέμα η ομοφωνία του Συμβουλίου. Πώ νομίζω ότι μπορέσουν, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τέτοιε ομάδε. Επίση, για το πακέτο τη Ευρωπόλ, θα ήθελα να σα παρακαλέσω θερμά, κύριε Υπουργέ, να κατανοήσετε ότι η ζωτικότητα τη Ευρωπόλ εξαρτάται από το κοινοβούλιο μα. Και είναι απαραίτητο να έρθουν το ταχύτερο δυνατό σε εμά οι εκθέσει Δία Δεμέρα και Άλμπρεχτ για τα θέματα τη Ευρωπόλ Για το Frontex, κύριε Υπουργέ, σε τι συνίσταται συντίστανται οι κατευθυντήρες γραμμές της ε, μεταρρύθμισής σας και τα 83 εκατομμύρια που αναφέρετε και σε σχέση με την τρομοκρατία πώς θα λειτουργήσει αυτό η Europol, το κέντρο συντονισμού. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά κάντε σας παρακαλώ ό,τι είναι δυνατόν ώστε να υπάρξει σωστή συνεργασία στην Ευρώπη. Και για το σύμφωνο ε, πληροφόρηση του Σέγγεν ο Κάλλος Κουέλιο, ο οποίος θα γνωρίζει καλύτερα τα θέματα αυτά και μπορεί να σας πληροφορήσει. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ασχοληθείτε, το είπατε ήδη για το έγκλημα στο κυβερνόχωρο, για τα θέματα του, της λεύκανσης χρημάτων και για τα θέματα σύντο. Ευχαριστώ. Σε δύο λεπτά δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την πληθώρα ερωτήσεων που μου έχουν θέσει. Θα ήθελα δύο ώρες για να μπορέσω να αντιμετωπίσω ενδελεχώς όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί. Γι' αυτό θα προσπαθήσω και ζητώ την επίοικια της ε, Προεδρίας να σας πω για το κόσι δεν έχουμε ακόμα καθορίσει ποιος θα είναι μέλος αυτής της ομάδος. Η προσωπική μου απλώς εντύπωση αυτή τη στιγμή είναι ότι το κόσι θα πρέπει να αποτελείται από τους ηγέτες των αστυνομιών των κρατών μελών και εγώ θα υποστήριζα ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να καταργήσουμε και την task force των αρχηγών των αστυνομίων που τελικά δεν έχει λειτουργήσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι το COS είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε μια λειτουργική συνεργασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ένα λειτουργικό όργανο, απλώς εγγυάται μιας καλύτερης λειτουργικής συνεργασίας και μιας ενότητας δράσης των θεσμικών οργάνων. Όπως είπατε, θέλουμε πράγματι να έχουμε ενιαίους συντονιστές για όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία και αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να μην δημιουργήσουμε ένα φορέα ο οποίος θα έχει υπερβολική γραφειοκρατία, όχι ένα όργανο το οποίο επικαλύπτεται με άλλους φορείς, αλλά να δημιουργήσουμε ένα φορέα ο οποίος θα έχει αρκετή ευθύνη των μελών του για να μπορέσει να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα αυτά, τα λειτουργικά αυτά. Και γι' αυτό πρέπει να έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Για τα θύματα της τρομοκρατίας δεν μπορώ παρά να είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σας σε σχέση με το θέμα αυτό βέβαια δεν είχα αρκετό χρόνο για να καλύψω όλα αυτά τα θέματα, αλλά σίγουρα η χώρα μας, η Ισπανία, έχει θυγεί ιδιαίτερα από τα θέματα της τρομοκρατίας. Έχω, την υποστήριξη, έχω πλήρη υποστήριξη προς τα θύματα της τρομοκρατίας και θα πράξω ό,τι είναι δυνατό ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να μείνει πάντα ζωντανή η μνήμη τους. Για το SWIFT, το PNR και τους αρωτές σώματος, το θέμα του SWIFT, αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τους Υπουργούς Εργασίας όχι η εργασία, συγγνώμη, η δικαιοσύνη διορθώνει ο κ. Υπουργό και επομένω δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στο δικό μου χώρο. Νομίζω ότι θα ήταν κάπω ανεύθυνο από τη δική μου πλευρά, εάν δεν σα έλεγα ποια είναι η δική μου άποψη ω Υπουργού Εσωτερικών. Εγώ κατανοώ απόλυτα τις διαφορές απόψεων που μπορεί να υπάρχουν, κατανοώ τις δυσκολίες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατανοώ επίσης προφανώς την διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισέλθει και αυτό στην ουσία του θέματος και να μπορέσει να αναλύσει σε βάθος αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Απλώς σας ζητώ να σκεφτείτε δύο πράγματα. Πρώτον, την χρησιμότητα του SWIFT και επομένως τη σημασία που έχει για τον αγώνα κατά του εγκλήματος, ιδίως κατά της τρομοκρατίας. Είναι μια χρησιμότητα πολύ μεγάλη που δεν πρέπει να την αποχωριστούμε για να εξασφαλίσουμε την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον αυτό το οποίο ήδη ζήτησε η Κομισιόν πριν από την Ισπανική Προεδρία αλλά και εδώ νιώθω υπεύθυνο, είναι το γεγονός ότι χρειάζονται εννέα μήνες μεταβατικού συστήματος ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει μια εικόνα για όλα αυτά και να καταλήξουμε μετά σε ένα οριστικό SWIFT όπου θα έχουν καλυφθεί όλες οι ανησυχίες, όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί. Και θα ήθελα εξάλλου να έχουμε μια συμφωνία με τους ε, εταίρους μας σε σχέση με τον αγώνα κατά του διεθνούς εγκλήματος και του οργανωμένου εγκλήματος που είναι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάνε μια δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή, μια ιδιαίτερα λεπτή στιγμή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αντίδρασή τους όταν έχουμε να λάβουμε αποφάσεις. Και πάλι σας λέω δεν είναι θέμα της άμεσης αρμοδιότητα, Θα ήθελα να σας ζητήσω να κατανοήσετε το λόγο για τον οποίο εμείς συναντηθήκαμε στο Τολέδο για να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτοί οι εννέα μήνες μεταβατικής περίοδου για το SWIFT με την κατανόηση ότι είναι μεταβατική και ότι στο οριστικό σύστημα θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο εξασφαλίζει και την ε, αντανάκλαση της ευαισθησίας και των φόβων, των λογικών φόβων των Ευρωπαίων πολιτών που θέλουν να είναι ασφαλισμένοι αλλά να έχουν και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή για το Passenger Name Record, για τα, τη συμφωνία αυτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ξέρετε, εμείς ως Υπουργοί Εσωτερικών θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να έχουμε μια συμφωνία για τα προσωπικά δεδομένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζουμε ότι από αυτή την άποψη είναι ουσιώδης και κεφαλαίωδης η ασφάλεια και έχουμε δεσμευτεί και πάλι με το Κοινοβούλιο για να δούμε ποια μέτρα, ποιοι έλεγχοι, ποιοι περιορισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται στο σύστημα αυτό για να εξασφαλίσουμε αυτή την πάρα πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας και να παραμείνει αυτή η ισορροπία στις παραμέτρους που έχει διατηρήσει, διατηρήσει η Ευρώπη σε όλο το παρελθόν της. Είναι τόσο λεπτή αυτή η ισορροπία, παρόλα αυτά εμείς την κρατάμε ζηλοτύπως γιατί είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ταυτότητας για του αρωτές πλήρου σώματο. Εγώ θα προτιμούσα να περιμένουμε τις τρεις αυτές εκθέσεις που εκπονεί η Κομισιόν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των σαρωτών πλήρου σώματος, το τι μπορούν να κάνουν το τι δεν μπορούν να κάνουν και επίσης θα, θα πρέπει να ελέγξουμε την συμβατότητά τους με τα ατομικά δικαιώματα, ιδίως τα, την ιδιωτική ζωή και επίσης την ενδεχόμενη επιρροή τους στην ε, υγεία των πολιτών. Όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία από τις τρεις εκθέσεις θα μπορέσουμε να έχουμε μια γαλήνια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα των σαρωτών πλήρου σώματος και θα μπορούμε να κάνουμε την κατάλληλη συζήτηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με τον κύριο Διάστε Μέρα, δεν έχω να προσθέσω κάτι για το Frontex εξάλλου. Η Κίνκα Κόνς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ισπανική Προεδρία είναι η πρώτη Προεδρία που λειτουργεί υπό το καθεστώς της συνθήκης της Λισαβόνας και με τη συνεργασία των δύο επόμενων ε, προεδρών που αποτελούν την Τρόικα, τη Βελγικής και τη Ουγγρική. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε του στόχου μα. Θα να κάνω ε, ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τι θεωρήσει. Καταρχά. νομίζω ότι σημειώνονται κάποια σημαντικότατα βήματα υπό την έννοια του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αναγνωρίζουν αυτόματα την αμοιβαία την, τις θεωρήσεις. Παρ' όλα αυτά γίνονται και βήματα προς τα πίσω, γιατί ο Καναδάς έχει ε, επανεισάγει την υποχρέωση θεωρήσεων για τους Τσέχους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η Ισπανική Προεδρία σκοπεύει να κάνει κάτι για αυτό το θέμα και αν ναι, τι. Τι σκοπεύει να κάνει για να εμποδίσει ούτω ώστε να υπάρχουν τέτοιου τύπου κινήσεις ε, όπως αυτή του ε, Καναδά. αυτή η υποχρέωση είχε καταργηθεί και τώρα επανεισήχθη για τους Τσέχους. Επίσης υπάρχουν σχέδια από Ισπανική Προεδρία για να υπάρξει διευκόλυνση των θεωρήσεων για τις ε, ε, χώρες της Νότια και Ανατολική Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Όπως ξέρετε και η πολιτική προξενικών θεωρήσεων δεν είναι αρμοδιότητα των Υπουργών Εσωτερικών και δικαιοσύνη, παρά το γεγονό ότι είναι γεγονό ότι γίνεται κάποια διαβούλευση μεταξύ μας σε σχέση με τις διευκολύνσεις για τα θέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά, για τις ε, θεωρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ξέρετε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ένα καθεστώς, ας το πούμε έτσι, μη αποδεκτό έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από προξενική θεώρηση και εμεί επιμένουμε να εφαρμοστεί και στις πέντε αυτέ χώρε το ίδιο καθεστώ όπω και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, μα φαίνεται απαράδεκτο να έχει επιβληθεί η υποχρέωση βίζα για τους πολίτες της Τσεχική Δημοκρατία στον Καναδά. Εμεί έκριναμε μια απόφαση στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών τον προηγούμενο Νοέμβριο, μια συμφωνία του Συμβουλίου των Υπουργών για να επιφορτήσουμε την Κομισιόν να εργαστεί κατεπηγόντως μαζί με τον Καναδά για να έρθει αυτό το οποίο εμεί θεωρούμε ότι είναι μια διάκριση εναντίον των πολιτών της Τσεχίας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τα εισαγωγικά σας λόγια. Καταρχάς, να χαιρετήσω την ε, επιλογή που έχει κάνει η Ισπανική Προεδρία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Παρ' όλα αυτά έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις για τα PNR και για το SWIFT. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα ένα ψήφισμα για τα PNR τον Νοέμβριο του 2008 και ζητούσε από το Συμβούλιο κάποιες εξηγήσει. Ουδέποτε λάβαμε απάντηση όμως. Νομίζω ότι είναι κάπως νωρίς να ξεκινάμε πάλι με το σχέδιο αυτή τη στιγμή που δεν μας έχουν δοθεί απαντήσεις όσον αφορά τώρα στο SWIFT υπογραμμίσατε την ε, χρησιμότητα του συστήματος αυτού των δεδομένων SWIFT. Εμείς όμως ακόμα αναμένουμε κάποιες πληροφορίες για τη χρησιμότητα αυτή και μάλιστα το θέσαμε αυτό, την, ε, το να λάβουμε τις πληροφορίες αυτές ως προϋπόθεση προκειμένου να ψηφίσουμε σε δύο εβδομάδες. Και τα μόνα έγγραφα τα οποία λάβαμε είναι τα πρωτόκολλα της συμφωνίας τα οποία μπορούμε μόνο να κοιτάξουμε σε ένα ασφαλέ δωμάτιο, σε μια ασφαλή αίθουσα και μόνο στο Συμβούλιο. Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι σωστή συνεργασία ανάμεσα σε δύο θεσμικά όργανα. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα, η συμφωνία με τις ΗΠΑ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου προσωρινά. Το Συμβούλιο περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή για να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σύμφωνη γνώμη του. Και ζητήσαμε επίσημα από το Συμβούλιο να αναβάλει τη θέση σε ισχύ και από ό,τι έμαθα δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα να ξέρω γιατί. Μας δίνουν μόνο πέντε μέρες και δεν μας δίνεται πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να λάβουμε τις αποφάσεις μας. Θεωρώ ότι δεν ξεκινάμε πολύ καλά στη συνεργασία στα πλαίσια της α, συνθήκης της Λισαβόνας. Και μια εντελώ διαφορετική ερώτηση τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη τα οποία δεν αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα του δικαστηρίου του Στρασβούργου, ιδίω όσον αφορά τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Και η Ισπανία επιβεβαίωσε ότι η ίδια συνάδει με τις αποφάσεις, με τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου. Θέλουμε να ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η δικιά σας άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω να σε ευχαριστήσω για, τα θέματα, για την υποστήριξή σας στα θέματα ισότητας των, των φύλων και μείωσης της βίας κατά των γυναικών. Για το PNR έχουμε μια προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ και με την Αυστραλία. Πρέπει να συζητηθεί αυτό με το Κοινοβούλιο σας, όπως πρέπει να συζητήσουμε και την, ζήτηση, την αίτηση των Υπουργών Εσωτερικών για τα περιεχόμενα του PNR. Θα πρέπει να συζητηθούν λοιπόν τα νέα στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν νομίζω εάν θέλουμε να έχουμε μια, ένα ευρωπαϊκό PNR, σίγουρα αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Δεν γνωρίζω πολύ καλά τις ε, συνήθειες ε, που έχετε, πώς ε, θα ψηφιστεί αυτό το προσωρινό SWIFT. Εκεί που θέλω να επιμείνω είναι ότι πρόκειται, όπως τονίσατε και εσείς, για ένα προσωρινό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει για εννέα μήνες. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα αυτό του SWIFT στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόκειται απλώς για να παρατείνουμε για λίγους μήνες ακόμα αυτήν την ε, συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Για να ξεπεράσουμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα μπορούμε να έχουμε όμως καλή συζήτηση, καλή εργασία. Αυτό το οποίο ζητώ από το Κοινοβούλιο είναι να αποδεχθεί αυτό το μεταβατικό διάστημα. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ και να χαιρετήσω την παρουσία σας στην Επιτροπή μας και θέλω να σταθώ σε τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ένα σημαντικό θέμα, όχι για να μας δώσετε απάντηση, για να πάρετε το μήνυμα και να το καταγράψετε. Για το θέμα του SWIFT είναι απαραίτητο να γνωρίζει το Συμβούλιο ότι η θέση που θα λάβουν για το θέμα αυτό θα θεσπίσει ένα προηγούμενο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το γνωρίζει το Συμβούλιο, δεν θα προχωρήσουμε στο ζήτημα αυτό μέχρι ότου υπάρξει μια απόφαση του Κοινοβουλίου, όχι μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στην ακολουθητέα διαδικασία. Είναι κάτι που είπαν και πολλοί προηγούμενοι ομιλητέ. Ο δεύτερο άξονα τη παρέμβασή μου έχει να κάνει με ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε και στο οποίο έχετε πιο άμεση ευθύνη. Έχει να κάνει με όλα τα θέματα τα οποία συνάπτονται με την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Και εδώ θέλω να εκφράσω τη λύπη μου. Γιατί πολλές φορές τα θέματα αυτά της ασφάλειας και της μετανάστευσης συγχέονται και συνενώνονται όταν είναι τελείως διαφορετικά θέματα σε πολλές περιπτώσεις. Και θέλω να υπογραμμίσω ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα κανονικό που βλέπουμε τις επιπτώσεις του κάθε μέρα στην καθημερινή διαχείριση της ε, μετανάστευσης. Δημιουργείται μια ψευδής ανασφάλιση, ανασφάλεια στον πληθυσμό και πολλές φορές συνδέεται με άλλα προβλήματα τα οποία είναι χωριστά, όπως το γεγονός ότι οι Δήμοι δεν έχουν αρκετά χρήματα για να αντιμετωπίσουν τα θέματα της μετανάστευσης. Επομένως το ερώτημά μου είναι το εξής. Από την άποψη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, η συμφωνία η οποία έχει ληφθεί μέχρι τώρα είναι μια συμφωνία που βασίζεται πάρα πολύ στην πτυχή της ασφάλειας. Σε μηχανισμ... Μας λείπουν ακόμα οι κατάλληλοι νομικοί μηχανισμοί. Επίσης, σε ό,τι αφορά την πολιτική παροχή ασύλου είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει αναγνώριση του προβλήματος αυτού ότι είναι δύσκολη απόδοση του ασύλου και επίσης σε σχέση με το θέμα της ε, συνεργασίας των αστυνομιών. Έχουμε σε ορισμένα κράτη σώματα αστυνομικά τα οποία είναι αποκεντρωμένα και όχι μονάχα εθνικά και επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτή η διάσταση. Ο κύριος Υπουργός καταγράφω προφανώς όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει και φυσικά ε, γνωρίζω σε σχέση με το θέμα SWIFT και ελπίζω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην αυριανή του παρουσία θα μπορέσει να δώσει μια ευρύτερη απάντηση στα θέματα αυτά που εγώ δεν μπορώ να σας δώσω γιατί δεν είναι πράγματι η αρμοδιότητά μου επί της ύλης για τα θέματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Σας έχω πει και προηγουμένως πώς θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά της μετανάστευσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Πιστεύω ότι αυτό αντανακλάται και στην συνθήκη και θεωρώ ότι αυτή η πολιτική πρέπει να έχει ένα οικουμενικό χαρακτήρα και να καλύψει τα τρία στοιχεία τα οποία βρίσκονται στη βάση του προβλήματος μετανάστευσης που είναι η ανάγκη να έχει η Ευρώπη μια νόμιμη μετανάστευση ώστε να υπάρχουν εργαζόμενοι και να υπάρχει η δυνατότητα να έρχονται άνθρωποι να εργαστούν στην Ευρώπη. Το θέμα λοιπόν της νόμιμης μετανάστευσης. Δεύτερον, την άλλη όψη του νομίσματος που είναι ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση απλώ κλείνοντα τα σύνορά μα γιατί πρέπει να συνεργαστούμε με τι χώρε διέλευση και προέλευση και μονάχα μπορούμε να συνεργαστούμε αν δίνουμε πραγματικέ δυνατότητε στου πολίτε των χωρών αυτών στην Ευρώπη και τρίτον είναι η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να εμπλακούν σε μια συνολική πολιτική. Μπορεί να είναι διαφορετική υπεύθυνη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του. Και κυρίω ο αγώνα κατά τη παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και του άλλου δύο παράγοντε. Εάν δεν υπάρξει κάτι δεν θα είναι επιτυχή. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πείσουμε τι χώρε προέλευση και διέλευση να μας βοηθήσουν και πρέπει να μας βοηθήσουν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί από εκεί, από την πηγή του φαινόμενου της παράνομης μετανάστευσης το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό όμως χωρίς μια βοήθεια προς τις χώρες αυτές για την ανάπτυξή τους και χωρίς δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία πρέπει να έχει η πολιτική μας και αυτά δεν έχουν μεγάλη σχέση με την κλασική σύλληψη της ε, ασφάλειας, γιατί η ασφάλεια έχει άλλες πτυχές πολλές φορές πιο πολιτικού χαρακτήρα. Υπήρξαν τα γεγονότα σε ορισμένου Δήμου τη Ισπανία, όπου υπήρξε και μια αναμόχλευση πολιτικών φόβων. Δεν πρέπει λοιπόν να το δούμε με ξενοφοβία το πρόβλημα αυτό, αλλά με λογική και διάλογο. Για το άσυλο δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν γνωρίζω το θέμα αυτό σε λεπτομέρεια και για τις αστυνομίες γνωρίζετε ποια είναι η θέση μου γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Έχουμε θαυμάσια συνεργασία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας με τις, πολυ... με τις αστυνομίες των ε, ομόσπονδων κρατών των αυτόνομων ε, περιφερειών, αν θέλετε, και αυτό απλώς θέλω να πω. Κύριο Στοβάρεσ. Κύριε Υπουργέ, στα πορτογαλικά μια ερώτηση, ή μάλλον δύο ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την ελευθερία διακίνησης. Πρώτα σε ό,τι αφορά το διατλαντικό χώρο και δεύτερο στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο κύριο Υπουργό αναφέρθηκε στην ενισχυμένη συνεργασία με τι ΗΠΑ στον αγώνα κατά τη τρομοκρατία και είναι προφανέ ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε κατανοούν ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την απειλή τη διεθνού τρομοκρατία είναι απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο. Αλλά είναι απαραίτητο και από την πλευρά των ΗΠΑ να έχουμε κάποια στοιχεία εμπιστοσύνη, ιδίω σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των επιβατών. υπάρχουν οι μαύροι κατάλογοι για τους Αμερικανούς πολίτες οι οποίες είναι υπό επανεξέταση, αλλά τίποτα δεν γίνεται για τους Ευρωπαίους επιβάτες. Δεν γίνεται καμιά προσπάθεια να εξεταστεί γιατί αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται στο, στη μαύρη λίστα των Αμερικανών ή αν θα πρέπει να φύγουν από αυτές τις λίστες. Δεύτερον, ελευθερία διακίνηση στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή είναι μια ουσιαστική ελευθερία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να μείνει όμως σε αφηρημένο επίπεδο. Πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη ελευθερία και έχει να κάνει και με το θέμα της επανένωσης οικογενειών και έχει να κάνει επίσης και με το θέμα της, ε, των ζευγαριών του ιδίου φύλου που μπορεί να είναι αποδεκτή η ένωση του σε μια χώρα αλλά όχι στην γειτονική χώρα. Θα πρέπει λοιπόν επομένως να γίνει κάτι σε αυτό το θέμα ή θα πρέπει να περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν αναγνωριστές αυτές οι ελευθερίες μέσα από τις, από τις εκλεγμένες συνελεύσεις των κρατών μελών, αλλά μόνο μετά από δικαστικές διαδικασίες. Για το SWIFT, εγώ θέλω να σας πω κύριε Υπουργέ, ότι δεν πρόκειται για μια μεταβατική συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία θα δημιουργήσει, θα θεσπίσει πρακτικές οι οποίες θα συνεχίσουν ως προηγούμενο και στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και πέντε χρόνια και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να μιλάμε για προσωρινές λύσεις. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε μέτρα τα οποία κινδυνεύουν να είναι μία αντιστρεπτά. Ευχαριστώ κύριος Υπουργός. Πάλι σύντομα σας ε, ζητώ συγγνώμη γιατί με τη χαρά μου που μιλήσατε στα Ισπανικά, έχασα λιγάκι από την μετάφραση. Αυτά που είπατε στα Πορτογαλικά, προσπάθησα να σα ακούσω και στα Πορτογαλικά και ίσω δεν ακολούθησα όλα αυτά τα οποία είπατε. Στα θέματα τη συνεργασία με τι ΗΠΑ, κατανοώ απόλυτα την ουσία τη ερώτησή σα. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα ισότητα να ζητάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πολίτες της Ευρώπης την ίδια μεταχείριση που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτείων. Μία αμοιβαιότητα μεταχείρισης. Ό,τι μας ζητούν οι, οι Αμερικανοί θα πρέπει να το ζητάμε και εμείς από αυτούς. Και φυσικά συμφώνω για το θέμα αυτό. Αν μου επιτρέπετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα υπάρχει μια συζήτηση για το να αναθεωρηθούν οι μαύρες λίστες επιβατών Αμερικανών και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να απαιτήσουμε από τους Αμερικανούς η αναθεώρηση αυτή να αφορά και τους Ευρωπαίους πολίτες και να υπάρχει μια δυνατότητα έφεσης αν για λανθασμένους λόγους έχουν συμπεριληφθεί σε αυτές τις λίστες. Ναι, πράγματι γίνεται αυτή η αναθεώρηση, έχετε δίκιο. Γιατί προσπαθούν να δούμε τι ακριβώς πήγε στραβά στην υποτιθέμενη αυτή απόπειρα του αεροπλάνου που πήγαινε στο Detroit. Μάλλον αυτό το οποίο έλειπε, αυτό το οποίο αστόχησε ήταν η δυνατότητα να συνδυαστούν διάφορες πηγές πληροφοριών. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μετά από συζήτηση στο Συμβούλιο θα πρέπει να τεθεί υπόψη των Αμερικανών. Μου είπατε επίσης το θέμα της ελευθερίας διακίνησης σε σχέση με τα <clears throat> ζευγάρια ιδίου φύλου και το οικογενειακό δίκαιο. Προφανώς ποικίλει το οικογενειακό δίκαιο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αυτό το οποίο ισχύει στη χώρα μου δεν είναι δεκτό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει, είναι σαφώς η ελευθερία διακίνησης χωρίς καμία διάκριση. Και το τελευταίο ερώτημά σας νομίζω ότι αναφερ, αναφερθήκατε στο SWIFT, αν κατάλαβα καλά. Δεν ζητούμε τίποτα το οποίο είναι χωρίς επιστροφή, μη αντιστρεπτό. Απλώς ζητάμε την παράταση του συστήματος που ισχύει όλα αυτά τα χρόνια με τη δέσμευση ότι μέσα σε 9 μήνες θα τα αναθεωρήσουμε και θα καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι οριστικό και θα περιλαμβάνει όλες τις λογικές διασφαλίσεις που μπορεί να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις διασφαλίσεις λοιπόν αυτές και την απαραίτητη διαφάνεια να μπορέσουμε να βρούμε αυτή την ισορροπία που πάντα υποστηρίζουμε και εμείς ήδη μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Ο κύριος Μπορκέτσιο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για κάποια σημεία που είπατε, για την καταπολέμηση της Ισλαμικής, Ισλαμικής τρομοκρατίας που είναι μεγάλος κίνδυνος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Έρασμους για τις αστυνομίες είναι ένα από τα θέματα όπου η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει περισσότερα. Εκεί όπου ήσασταν αρκετά γενικόλογος είναι το γενικό θέμα της μετανάστευσης. Για σας, τι σημαίνει καταπολέμηση της ε, λαθρομετανάστευσης. Τι είναι αυτό. Πρόσφατα ο πρόεδρος Σαρκοζή έλαβε θέση για αυτό το θέμα ένα ε, πολιτικό στην Ευρώπη που επιτέλου θα παίξει από τα δόντια. Είπε ότι δεν πρέπει να διατρέξουμε τον κίνδυνο να γίνουμε, είπε εκείνο, ε, αυτό που έγινε η Ιταλία. Εγώ το διορθώνω λιγάκι αυτό που είπε ο κ. Σαρκοζή. Θα είχαμε γίνει στην Ιταλία αυτό που είπε ο κ. Σαρκοζή, αν ο κ. Μαρόν δεν έπαιρνε αυτά τα μέτρα που πήρε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα στην Ιταλία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το συζητάμε συνέχεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να μα ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Ποια είναι η ευρωπαϊκή πολιτική που προτείνεται συγκεκριμένα για να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση. Μπορείτε να μας πείτε. Κύριε Υπουργέ. Προσπάθησα να το εξηγήσω προηγουμένως, θα το κάνω και τώρα πάλι. Νομίζω ότι έναντι της ε, παράνομης μετανάστευσης προφανώς θα πρέπει να γίνει ο αγώνας στα σύνορά μας, είτε είναι χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια. Τα πιο δύσκολα σύνορα είναι τα θάλασσια, γι' αυτό εστιάζεται ένα μεγάλο μέρο στι προσπάθειε τη Frontex από τη θάλασσα. Στη θάλασσα, βέβαια, τα σύνορα τα θαλάσσια έχουν και μια άλλη πτυχή που είναι πάρα πολύ σημαντική, την ανθρωπιστική διάσταση, γιατί κινδυνεύουν να πνιγούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται. Αλλά για τα σύνορά μα είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μπαίνουν μέσα από τα σύνορά μα άτομα χωρί <clears throat> χωρίς έγγραφα να έχουμε ασφαλή σύνορα. Δεν μπορούμε όμω να λησμονήσουμε τη συνεργασία με τι τρίτε χώρε που έχει δύο σημαντικέ πτυχέ, την πολιτική επαναπατρισμού και τον αγώνα κατά τη παράνομη μετανάστευσης στις χώρες διέλευσης ή στι χώρε προέλευση των μεταναστών. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, το οποίο δείχνει πραγματικά ποιε είναι οι πρακτικές που πρέπει να διατηρήσει η Ευρώπη. Η Ισπανία με τη Σενεγάλη, παραδείγματο Η Ισπανία είχε ένα πρόβλημα με τη Σενεγάλη τεράστιο το 2006 γιατί ήρθαν πάνω από 20.000 Σενεγαλέζοι στη χώρα μας. Ξεκινήσαμε μια πολιτική με τη Σενεγάλη που είχε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, δώσαμε στη Σενεγάλη τη δυνατότητα να έρχονται οι Σενεγαλέζοι και να εργάζονται σε ορισμένε περιοχέ που χρειαζόταν εργαζομένου η Ισπανία. Δεύτερον, του βοηθήσαμε να ελέγξουν τα σύνορά του. Και τρίτον, ξεκινήσαμε προγράμματα συνεργασία για να ευνοήσουμε την ανάπτυξη τη Σενεγάλη. Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να συμμετέχει και η Σενεγάλη στον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης και μια τέτοια αντιμετώπιση ήταν η καλύτερη δυνατή. Και αυτό πρέπει να γίνει με όλες τις χώρες από τις οποίες έρχονται μεταναστευτικά ρεύματα να δεσμευτούν, να έχουν αυτή τη συνεργασία και τις, ε, <clears throat> τους επαναπατρισμούς έναντι της συνεργασίας για την ανάπτυξη, τότε σταματά αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα. Μπήκαν Σενεγαλές πια νόμιμα στην Ισπανία, αλλά όχι παράνομα πια. Έχουμε καλύψει τον πρώτο γύρο με την μέθοδο DONT, δηλαδή ένα ομιλητή από κάθε πολιτική οικογένεια που αντιπροσωπεύονται στην Επιτροπή μα. Δύο λεπτά ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση. Είναι απαραίτητο όμω ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον στην, από την παρουσία του κ. Υπουργού και είναι τεράστιο ο κατάλογο, είναι μεγάλο ο κατάλογο των μελών που θέλουν να λάβουν το λόγο. Αν συνεχίσουμε έτσι, πολλοί δεν θα προλάβουν να λάβουν το λόγο. Προτείνω επομένω να αλλάξουμε μέθοδο για να δώσουμε το μεγαλύτερο δυνατό στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό βουνευτών να λάβουν το λόγο. Σας προτείνω ο καθένας να μιλάει για ένα λεπτό και να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, ώστε στη συνέχεια συνολικά ο κύριος υπουργό να μπορέσει να απαντήσει ομαδικά στους βουλευτές, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να ικανοποιήσουμε το μεγαλύτερο αριθμό αυτών οι οποίοι θα λάβουν το... Η Βαρονίσα Λάτφορντ. Η κυρία Ινβέλτ μίλησε όμως ως αντιπρόεδρος, έτσι δεν είναι. Ακολουθήθηκε η, η διαδικασία... Όχι, όχι, μίλησε εξ ονόματος των α, φιλελευθέρων. Πρώτη εξ ονόματος των φιλελευθέρων μίλησε η κυρία Ινβέλτ, το διευκρινίζω. Ένα λεπτό καθένας πλέον και θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός με διαχείριση του χρόνου. Ο κύριος Κουέγιου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, άκουσα με μεγάλη ευχαριστήση την παρέμβασή σας και αυτά που αναφέρατε στο σχέδιο αυτό, το οποίο έχει σαν στόχο να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες, με παράλληλη ενίσχυση των ελευθεριών τους. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειες της Ισπανικής Προεδρίας. Εγώ <clears throat> ανησυχώ για την ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων με παράλληλη εξασφάλιση της ελευθερίας διακίνησης μέσα στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε στο σύστημα πληροφορίας του Schengen, το ΣΥΣ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σας θα μπορέσετε να πάρετε μια απόφαση για το ΣΥΣ2 και αν το ΣΥΣ2 δεν λειτουργήσει σωστά, έχετε μια, ε, οδό, μια εναλλακτική οδό σε σχέση με την, τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ κύριε Κουέλιο. Ο κύριος Ρομέρο Λόπεθ, η κυρία Λόπεθ μάλλον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να υποδεχθώ τον Υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας και θα είμαι σύντομη. Κύριε Υπουργέ, διαπιστώνουμε ότι ο συντονισμό των διοκτικών αρχών, δικαστικών και αστυνομικών δεν επαρκεί ενώπιον των συνολικών απειλών που έχουμε. Εξάλλου, η συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί κατά ανάγκη και ένα ευρύτερο χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Και πρέπει να αντιμετωπιστούμε την τρομοκρατία μέσα στο κράτος του δικαίου. Και είμαστε επιπλεγμένοι και στην διατλαντική συνεργασία, όπου υπάρχει λόγω ακριβώ τη τρομοκρατία η έλλειψη εγγυήσεων όπω το αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Είναι δυνατόν αυτό ο συντονισμό των δικαστικών και αστυνομικών δυνάμεων να μπορέσει να οδηγήσει σε μια κοινή στρατηγική, να δημιουργήσουμε ένα θεσμό, μια επιτροπή, ένα όργανο το οποίο να συνδυάζει την αποτελεσματικότητα σε δικαστικό και αστυνομικό επίπεδο, ακόμα και στο οικονομικό επίπεδο. Ευχαριστώ η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Την ίδια ερώτηση θα κάνω σε εσά που έκανα στην κυρία Μάλστρομ στην ακρόασή τη. Μου δώσε θετική απάντηση. Δηλαδή, συμφωνούσε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο κατάλογος των μέσων που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή δεδομένων και για την γενική επιτήρηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικά στις διατλαντικές ε, σχέσεις. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν υποβληθεί πάρα πολλές προτάσεις ε, τις οποίες έχουμε απορρίψει, δεν έχουμε συμφωνήσει, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουμε, δεν υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Πότε θα έχουμε πλέον αρκετά δεδομένα πότε θα φτάσουμε στον τελικό μας στόχο, πότε θα πούμε ότι έχουμε πλέον αρκετές πληροφορίες για τους ανθρώπους, δεν χρειαζόμαστε άλλες πληροφορίες, αυτό που χρειάζεται πλέον είναι να συνδέσουμε τα στοιχεία μεταξύ τους και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Άκουσα πάρα πολλά σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και για την ανάγκη να υπάρξουν μέτρα ασφαλείας, εγώ θα χαιρόμουν αν το Συμβούλιο υποστήριζε καλύτερα αυτή την ανάγκη με αξιολογήσεις και με πραγματικά στοιχεία και αν μας τα έδινε αυτά τα στοιχεία τακτικά υπόψη μας. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε εμείς σαν νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση και επίσης αυτό το οποίο θα ήθελα να έχω από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια πιο νυφάλια <clears throat> αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά, όπου υπάρχει λιγότερη αναμόχλευση φόβων για τρομοκρατικές επιθέσεις και να υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση σε αυτό το οποίο πράγματι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε που είναι η εγκληματικότητα. Έχω ακούσει πολύ λίγα πράγματα από εσά για το πώς θέλετε να μειώσετε την εγκληματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς πέρα από τα μέτρα ασφαλείας θα αντιμετωπίσετε και την εγκληματικότητα. Ο κύριος Μπουσούτελ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθούμε πάλι στο ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης. Βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει οι διαδρομές, μάλλον που ακολουθούνται στην ε, παράνομη μετανάστευση. 30.000 στο παρελθόν είχαμε στη Λαμπεδούσα πέρυσι, αυξήθηκαν οι αριθμοί αυτοί στην Ελλάδα και πέρυσι την Παρασκευή έφτασαν παράνομοι μετανάστες στην ε, Κορσική. Αλλάζουν λοιπόν οι διαδρομές της παράνομης μετανάστευσης, πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι ε, τα εγκληματικά δίκτυα ουσιαστικά μας έχουν ξεπεράσει την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και ότι ε, η προστασία των εξωτερικών συνόρων θα πρέπει πραγματικά να είναι μια κοινή ανησυχία. Ποια είναι η άποψη της Ισπανικής Προεδρίας και τι προτίθεται να κάνει κυρία Ζίπελ. Μια ρητορική, αν θέλετε, έκφραση για το SWIFT. Εδώ και 8 χρόνια ζητάμε από τους Αμερικανούς να μάθουμε και δεν έχουμε πάρει καμία απολύτως απάντηση για όλα αυτά. Αυτό είναι εύγλωτο και από μόνο του μας δίνει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι σημαντικό για τα θέματα ασφάλειας να έχουμε μια στρατηγική, αλλά εδώ θέλω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα ότι πολλές φορές ακόμα και μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν μορφές εγκληματικότητας να μπορούν να μιλούν για τα θέματα αυτά. Όχι μόνο χανέοι που έρχονται από μετανάστευση, αλλά και αυτόχθονες πολλές φορές κάνουν δηλώσεις οι οποίες είναι απολογία της τρομοκρατίας. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στην ε, αντιμετώπιση των νέων. Ο κ. Μπιλμπάου. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ για όλες τις εξηγήσεις που μου δώσατε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο εξάμεινο σας. Μιλήσατε για την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών αστυνομικών δυνάμεων, να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σας θέσω το ερώτημα. Γιατί μέσα στην επιχειρηματολογία σας δεν έχετε ενσωματώσει πλήρως το πρωτόκολλο Σέγγεν τις, ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της χώρας των Βάσκων και η όπου η αστυνομία της χώρας των Βάσκων πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα όπως και η εθνική αστυνομία. Λοιπόν, με το να την αφήνετε έξω από το κύκλωμα αφ, μειώνεται την ασφάλεια αυτής της περιοχής και οδηγείται σε κατασπατάληση πόρων. Επίσης θα ήθελα στο πρωτόκολλο της Στοχόλμης να συμπεριλάβουμε μια τροπολογία που να αναφέρεται στα θύματα της τρομοκρατίας. Να υπάρξει μια ευρωπαϊκή χάρτα για τα θύματα της τρομοκρατίας ή όχι και ποια είναι τα θύματα τα οποία κατά την άποψή σας θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτή τη χάρτα, αν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εμπειρία των ε, εθνικών κρατών και την εμπειρία των ενώσεων των θυμάτων. Κύριος Μπόντς. Uh, uh, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ αναφερθήκατε σε μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση. Αν εγκριθεί η πολιτική αυτή, τότε θα ακυρώσει αστικά τις υποσχέσεις των πολιτικών αυτών από τα κράτη-μέλη που θέλουν να θέσουν τους δικούς τους περιορισμούς στην, στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Αναφέρουμε σε πολιτικούς που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπούν κράτη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Κίνκα Υπουργέ. Πάτα, Κύριε Υπουργέ, είμαι πολύ ικανοποιημένη για το κοινό πρόγραμμα που ανα, ε, εκπονήσατε μαζί με τους ε, Βέλγους και τους Σούγκρους. Νομίζω ότι αυτό ε, αποτελεί μια εγγύηση ότι μακροπρόθεσμα θα υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις ε, που για τις οποίες μιλάει και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Χαίρομαι επίσης που μιλήσατε για τη στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια και για τα εξωτερικά σύνορα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αλλά είναι πολύ σημαντική, αλλά και η καταπολέμηση τη οικιακή βία γενικότερα είναι πολύ σημαντική, στην οποία αναφερθήκατε. Νομίζω πρέπει να μιλήσουμε και για την προστασία των ανηλίκων. Ε, περιμένουμε συγκεκριμένε δράσει ε, και για την ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Επίσης, ε, για, ε, για την καταπολέμηση της βίας κατά των ανηλίκων. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ε, καταρχάς θέλω να σας χαιρετήσω, να χαιρετήσω το χαρακτηρισμό που κάνατε για το εξάμεινο αυτό, εξάμεινο για την καταπολέμηση της βίας γενικά. Ε, μία ερώτηση που την ανέφερε και η κυρία Γκάλ. Μεταξύ των προτεραιοτήτων σας, ή σκοπεύετε να ασχοληθείτε και συγκεκριμένα νομοθετικά ε, με την εκμετάλλευση, τη σεξουαλική εκμετάλλευση των υλίκων και την παιδοπορνογραφία στο ίντερνετ. Δεύτερον, μία πρόταση για το άσυλο. Νομίζετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα που προβλέπουν επιμερισμό των υποχρεώσεων μεταξύ όλων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις ε, ευθύνες τους. Δηλαδή, τι εννοώ, να προβλέψουμε μέτρα υποχρεωτικής επανεγκατάστασης. Αυτό για να αποφύγουμε ούτως ώστε κάποια κράτη-μέλη ε, φέρουν μόνα τους το βάρος που προκύπτει από την υποδοχή των προσφύγων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε στην επιτυχή σας συνεργασία με τη Σενεγάλη για να μπορέσει να ανακοπεί το ρεύμα παράνομης μετανάστευσης. πώς έγινε ο έλεγχος αυτής της ε, ε συμφωνίας. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των σχέσεων σας με το Μαρόκο χρειάστηκε κάποια άτομα να επαναπατριστούν. Πώς λοιπόν έχει αναπτυχθεί η συνεργασία σας με χώρες όπως το Μαρόκο, αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στην Τενερίφη και σε άλλους τόπους κράτησης και πώς αντιμετωπίζετε τις προσπάθειες να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να γίνεται με κοινό τρόπο αυτή η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και να μην αφήνονται χώρες όπως η Μάλτα στην τύχη της που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ένα τόσο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα παρά τη θέλησή της. Ο κύριος Χιμένες, η κυρία Χιμένες. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι απαντήσατε και στα ερωτήματα του κυρίου Ντία Δεμέρα και επίσης για το γεγονός ότι έχετε αναγνωρίσει τη δέσμευση της Ισπανίας σε σχέση με τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι είναι πραγματικά απαραίτητο να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη αυτών των θυμάτων, γιατί είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που έχουμε για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο. Και πρόκειται για τη χάρτα αυτή ευρωπαϊκών δικαιωμάτων για τα θύματα της τρομοκρατίας που ανέφερε ο κ. Διάστη μέρα. Αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό το οποίο θέλω εγώ προσωπικά να επιτευχθεί είναι να υπάρξει η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων και το δικαίωμά του να τύχουν να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης. Γιατί μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιστρέφονται από την τρομοκρατία είναι πολύ δύσκολο να έχουν μια δικαίωση σε δικαστικό επίπεδο. Επομένως θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα υπάρξει η επίτευξη αυτής της χάρτας δικαιωμάτων των θυμάτων και τι θα κάνετε για να επιτύχετε την προσχώρηση και των άλλων κρατών μελών, ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να προσβλέπουμε ότι θα έχουμε χάρη στις προσπάθειες της Ισπανικής Προεδρίας για να γίνει πραγματικότητα αυτή η χάρτα. Ευχαριστώ. Κύριε Κοτσέτα. Κύριε Κοτσέτα. Κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τις προτεραιότητες που μας αναφέρατε και κυρίως ε, για κάτι σημαντικό που είπατε. Ε, κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν το έχουμε συζητήσει αρκετά στην ε, σημερινή μας συζήτηση. Το θέμα της του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Συχνά μιλάμε για την τρομοκρατία, πολύ συχνά μιλάμε για τα θύματα της τρομοκρατίας. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω στους βουλευτές ότι σε αυτή την αίθουσα υπάρχει ο, η, αδερφή ενός δικαστή, η Ρίτα Μπορσελίνο, ο οποίος σκοτώθηκε από τη μαφία, ε, έγινε κοιμάς από μια βόμβα ε, της μαφίας. Ε, θα ήθελα κύριε Υπουργέ να δείξετε μεγαλύτερη ευαισθησία για το θέμα αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για τα θύματα της τρομοκρατίας, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματο από δίπλα. Όταν μιλάμε για του μάρτυρε που πάνε στα δικαστήρια, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για του μάρτυρε που πάνε στα δικαστήρια για να ε, μιλήσουν εναντίον του οργανωμένου εγκλήματο. Επίση, θα ήθελα να μιλήσουμε για την προστασία των θυμάτων, των μαρτύρων, όλων όσων εμπλέκονται. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη ε, αδιαφορία στο εσωτερικό τη Ευρώπη. Ε, σας ευχαριστώ που θέσατε αυτά τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Κυρία Πλίνκεβιτσιούτε. E, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανάμεσα στις προτεραιότητες αναφερθήκατε στην καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Δεν έγινε όμως κάποια αναφορά στην εμπορία ανθρώπων. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί τμήμα της βίας κατά των γυναικών, γιατί πολύ συχνά είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια που πολλούνται σαν σκλάβοι. Και το φαινόμενο αυτό δεν ελέγχεται αυτή τη στιγμή και ούτε προβλέπονται κυρώσεις. Οι γυναίκες και τα κορίτσια πολλούνται έρχονται από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις φέρνουν εδώ και συνέχεια πραγματικά τις ε, πουλάνε από τη μία χώρα στην άλλη. Πιστεύετε ότι ε, υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου από τον ένα μέλος στο άλλο. Θα λέγατε ότι οι αστυνομικές αρχές των κρατών μελών είναι σε θέση να συνεργαστούν επαρκώς και τι πρόκειται να κάνει η Ισπανία για το φαινόμενο αυτό. Έχω ακούσει πάνω από 15 λεπτά ερωτήσεων που εκφράζουν τις ανησυχίες και τις αβεβαιότητες των μελών της Επιτροπής μας. Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι όλα αυτά τα έχει καταγράψει ο κύριος Υπουργό, αλλά δεν μπορείτε να ελπίζετε ότι θα μπορέσει να δώσει μια λεπτομεριακή απάντηση. Είναι η τελευταία λοιπόν απάντηση του κύριου Υπουργού και νομίζω ότι θέλουμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε για αυτά που μας είπατε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποτέ μου δεν κατάφερα να καταγράψω τα ονόματα όλων των κοινοβουλευτικών που έλαβαν το λόγο γιατί δεν τους γνωρίζω ακόμα. Πρέπει να με βοηθήσετε και έχω <laughs> τελικά και πολύ, κακή, ε, πολύ κακογραφικό χαρακτήρα για το θέμα του συστήματος πληροφόρησης του Schengen. Αυτή τη στιγμή προχωρούμε σε μια αξιολόγηση του SIS2, της λειτουργίας του. Αν είναι θετικό ο απολογισμός, τότε τον Ιούνιο θα τεθεί σε λειτουργία. Αν είναι θετική η αξιολόγηση. Αν οποιαδήποτε από τι δύο αξιολογήσει είναι αρνητική, το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα σκεφτούν για δύο μήνε για το πρακτέο. Αν θα προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε το ΣΥΣ2 ή αν θα πρέπει να ενισχύσουμε το ήδη υπάρχον σύστημα, το ΣΥΣ1. Ακόμα και σήμερα, νομίζω χθες ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης. Εγώ προφανώς δεσμεύομαι να πληροφορήσω το Κοινοβούλιο για τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν και σίγουρα εδώ στον τομέα αυτό η πρωτοβουλία ξεκινάει από την Κομισιόν. Για το θέμα της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής, το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Ρομέρο, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέε μεγάλε, μεγαλόσχημε δομέ. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο αυτέ τι δομέ που έχουμε ήδη τώρα. Νομίζω ότι προς το παρόν η πληροφορία λειτουργεί με μεγάλη ευκολία για θέματα όπως αυτά της τρομοκρατίας και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μοιραστούμε περισσότερο, όπως δείχνουν τα πρόσφατα γεγονότα, να μοιραστούμε τις πληροφορίες και την ανάλυση των πληροφοριών αυτών, τα στοιχεία που συλλέγουν οι μυστικές υπηρεσίες και να κατατήσουν μια στρατηγική βάση αυτών. Να έρθουμε λοιπόν σε επαφή και με τους ε, ομολόγους μας στις οντότητες που αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία για να μπορούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να κρατήσω το όνομά σας. Πολλές φορές Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε ποιες από αυτές τις πληροφορίες είναι πράγματι χρήσιμες. Δηλαδή να περάσουμε από την απλή συλλογή πληροφοριών στην ενδελεχή και ευφυή ανάλυση τους. Για την εγκληματικότητα, αυτό είναι κάτι που απασχόλησε πάρα πολλού βουλευτέ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι στα θέματα ασφάλεια οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τους κοινού κινδύνους. Είναι γεγονό ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών, την ανασφάλειά τους, αλλά πολλά από αυτά καλύπτονται σε επίπεδο κρατών και ή αυτόνομων περιοχών ή αποκεντρωμένων μονάδων ακόμα και τοπικό επίπεδο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι πορτοφολάδες δημιουργούν την εντύπωση της ανασφάλειας στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά δεν μπορεί η ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει τους λαχανάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός όταν πρόκειται για μια οργανωμένη δραστηριότητα. Επίσης, πολλές φορές μπορεί πίσω από την κλοπή αυτοκινήτων να κρύβεται μια ομάδα οργανωμένη σε εγκληματικότητα σε διεθνικό επίπεδο. Τότε μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί όμως να παρέμβει σε όλα τα επίπεδα όταν πρόκειται για μικρού κλίματος έγκλημα τοπικού χαρακτήρα. Αυτό εναπόκειται στις εθνικές αρχές. Αλλά αυτό το οποίο λέτε ότι πέραν τη τρομοκρατία που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα πολλά τα οποία απασχολούν του πολίτε και τα οποία έχουν ακόμα περισσότερη επίπτωση στο αίσθημά του τη ε, προσωπική ασφάλεια ή ανασφάλεια, πρέπει να σα πω έχετε μεγάλο δίκιο και πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ περισσότερο από την τρομοκρατία και όλα αυτά τα θέματα τα οποία δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλεια. Χωρί να λησμονήσουμε την τρομοκρατία. Είναι γεγονό ότι όλοι οι ανθρώποι είναι επιλύσμονες και το Detroit ήταν έκρουσε τον κόδωνα κινδύνου για τα θέματα της τρομοκρατίας όπου η μνήμη μας είχε ήδη αρχίζει να χάνεται και θα πρέπει να δούμε ποιο κίνδυνο επικρέμαται αυτή τη στιγμή ενώπιόν μα, αυτό που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν είναι μεγαλύτερο ο κίνδυνο τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μεγαλύτερο ο κίνδυνο τώρα από ό,τι στο παρελθόν και επομένω πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλεία μα. Μιλήσατε για τη Μάλτα και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα τη Μα, της ε, Μάλτας, τα θέματα αυτά της Κορσίκης και το πλοίο με τη Γαλλία. Ξέρω ότι αλλάζουν συνέχεια οι διάβλοι της μαφίας. Τι, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αλλάζουν οι διάβλοι. Πρέπει να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας. Και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι οι χώρες διέλευσης για την ε, παράνομη μετανάστευση παραγωγής χάρη, πρέπει να σκεφτούμε και τις άλλες εναλλακτικές χώρες οι οποίες μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Και η γεωγραφία της Μεσογείου είναι σαφής. Αν υπάρξει μεγάλη αυστηρότητα στο, μεταξύ Ισπανίας και Βόρειας ε, Αφρικής, στη συνέχεια θα μετακομπιστεί αυτή η διαδραστηριότητα αλλού. Αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας και Λιβύης, πολλοί θα προσπαθήσουν να φύγουν από άλλες πλευρές στην Ανατολική Μεσόγειο, χάρη. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ευκαινησία για τις μαφίες λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων. Αυτό το οποίο όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι η ανάγκη να συνεργαστούμε με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα, όπως σας είπα προηγουμένως, να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τις χώρες αυτές και να τις βοηθήσουμε στην αναπτύξή τους. Αυτό είναι το ουσιώδες και να τους προσφέρουμε εναλλακτικέ λύσεις. Δεν μπορούμε σε Ευρώπη να σου λέμε όχι, όχι, να μείνετε απ' έξω. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους και να τους βοηθήσουμε για να έχουμε μια επιτυχή πολιτική. Συμφωνώ απόλυτα επίση με την ανάγκη πρόληψη. Μιλήσατε για την βία των νέων και το γεγονό ότι υπάρχουν ε, αυτοί οι οποίοι αναμοχλεύουν τη βία των νέων, ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση και σεμινάρια κατά τη ε, νεανική εγκληματικότητα, η οποία αυτή τη στιγμή κατεβαίνει στου εφήβου, ε, στα, στα μικρά παιδιά που έχουν μια όλο και βία αντιμετώπιση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ασφάλειας, αλλά περισσότερο σε επίπεδο ε, εκπαίδευσης. Η αστυνομία στη χώρα των Βάσκων είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για τη χώρα των Βάσκων, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι η συνεργασία μεταξύ της βασικής αστυνομίας και των Ισπανική αστυνομία και των άλλων αστυνομίων είναι όλο και καλύτερη. Βελτιώνουμε συνέχεια τον τρόπο συνεργασία. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να μπορέσει να προχωρήσει με ανεξαρτησία όλων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτά μπορούν να βοηθήσουν να υπάρχει μια επιτυχία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Για τα θύματα της τρομοκρατίας, εγώ υποστηρίζω το να υπάρχει μια χάρτα για τα θύματα της τρομοκρατίας, το υποστηρίζω όπως είπα και στον κύριο Διαστεμέρα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για κάτι το οποίο ενδιαφέρει τόσο πολύ και αγγίζει την ευαισθησία όλων των Ευρωπαίων. Είτε οι χώρε μα έχουν εσωτερική τρομοκρατία, είτε δεν έχει. Νομίζω ότι είναι ένα θεμελιώδε ζήτημα όπου πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και φυσικά οι χώρες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την τρομοκρατία και είναι πολλές μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα η εμπειρία των χωρών αυτών. Αναφέρθηκε το θέμα της υποχρεωτικής μετεγκατάστασης στην περίπτωση της Μάλτας. Εμείς έχουμε ένα εθελοντικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, όχι ένα υποχρεωτικό. Σίγουρα το πρόγραμμα της Στοκχόλμης έχει σαν στόχο να επισημοποιήσει τα συστήματα αλληλεγγύης. Βέβαια, αυτό δεν είναι απλό, γιατί υπάρχουν πολλέ χώρε οι οποίε βλέπουν από μεγάλη απόσταση το φαινόμενο τη παράνομη μετανάστευση. Η Προεδρία θα πρέπει να πει στι χώρε αυτέ, οι οποίε βρίσκονται σε μια απόσταση ασφαλεία, να καταλάβουν ότι υπάρχουν χώρε οι οποίε υφίστανται μια τεράστια μεταναστευτική πίεση, όπω η Μάλτα, η Ισπανία και η Ιταλία, και οι οποίε είναι τελικά τα σύνορα τη Ευρώπη τη ίδια. Μέσα από αυτήν την προοπτική, τα θέματα αυτά μετακίνηση μεταναστών θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε προγράμματα επισημοποιημένα για την εφαρμογή της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος Κροτσέτα στα εγκλήματα της μαφίας και κατανοώ απόλυτα ότι πρόκειται για μια πολύ καλά οργανωμένη μορφή εγκληματικότητος η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με τοπικά από όλε τι χώρε και επίση να τύχει συγκεκριμένη μνήμα ότι τα άτομα αυτά τα οποία αγωνίζονται κατά τη μαφία θα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη αναγνώριση. Και τέλο για το λαθρεμπόριο ανθρώπων δεν αναφέρθηκα σε αυτό ενδελεχώ. Όπω ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει σαν, σαν τίτλο Δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του λαθρεμπορίου ανθρώπων είναι κάτι το οποίο εκτελήσεται μεταξύ πολλών χωρών και υπάρχει και μια μη κυβερνητική οργάνωση στο Βέλγιο η οποία ασχολείται με αυτά. Είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ισπανία κτλ. Και υπάρχουν εργαλεία δράση τα οποία ξεκίνησαν την εποχή τη Σουηδική Προεδρία. Η Ισπανία είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα αυτό. Θα οργανώσει στι 4 Μαρτίου μια συνδιάσκεψη στη Μαδρίτη που οργανώνεται από την Ισπανική Προεδρία και ο στόχο μα είναι να μπορέσουμε να διαγράψουμε βασικέ γραμμέ ενό σχεδίου δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς μας απασχολεί το θέμα αυτό και είμαστε έτοιμοι στον τομέα αυτό να αγωνιστούμε κατά του λαθρεμπορίου ανθρωπίνων όντων, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Και τίποτα άλλο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας και για την προσοχή σας. Και προφανώς στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου θα επανέλθω να σας εξηγήσω τι πράττει η Ισπανική Προεδρία και ποια είναι η πρόοδος για τα θέματα αυτά που σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. συνάντηση ήταν πάρα πολύ πυκνή. Νομίζω ότι συμφωνούν και τα μέλη της Επιτροπής ότι ήταν και πολύ επικοδομητική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε όλους ιδιαιτέρως για τις εξηγήσεις σας. Ακούσατε τις ερωτήσεις των βουλευτών, κύριε Υπουργέ, και περιμένουμε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας ότι θα τα καταφέρει σε όλα τα μέτωπα στα οποία έχει θα δραστηριοποιηθεί. Σας ευχαριστούμε. Καθίστε σας παρακαλώ για να ξαναρχίσουμε. Καλησπέρα σε εκ νέου. Χαιρετίζουμε τον ε, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Εργασίας λοιπόν και Μετανάστασης της Ισπανικής Κυβέρνησης, ο οποίος θα παρουσιάσει στην Επιτροπή Εσωτερικών και Ελευθεριών το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας για τους επόμενους έξι μήνες ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Θα ακούσουμε την παρουσίαση του Υπουργού για 10 λεπτά και για να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο το χρόνο μας, θα ήθελα να κάνουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και παρεμβάσεων, κάθε μία δύο λεφτά, με βάση το σύνθεσή σύστημα DONT ε, και την εκπροσώπηση των πολιτικών ομάδων. Θα ακούσουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις ομαδοποιημένες από τον ε, Υπουργό και εν συνεχεία έναν δεύτερο γύρο με ερωτήσεις και απαντήσεις από τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον ε, λόγο και καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εμφανιστώ ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής, της Ισπανικής Συγγνώμη Προεδρίας στα θέματα της ε, νόμιμης μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Η έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας είναι μια ευκαιρία η Ευρώπη να γίνει πιο ανοιχτή, πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στους πολίτες. Οι αξίες αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν ουσιαστικά στο σχήμα μιας πολιτικής μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι ευρεία, θα είναι μόνιμη και θα είναι οικουμενική. Η ρύθμιση αυτή τη κοινή πολιτική μετανάστευση που εισάγεται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, κατά την άποψή μου, έχει τρία μεγάλα θετικά σημεία. Πρώτα απ' όλα, περιλαμβάνει μια ειδική νομική βάση για τον καθορισμό των δικαιωμάτων <clears throat> των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η νέα συνθήκη είναι σαφής σε σχέση με το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών που θα μπορούν να διαμένουν στο έδαφος τους. Τρίτον, η συνθήκη δημιουργεί μια νέα νομική βάση για κοινή δράση σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος τον οποίο αποδίδει η συνθήκη της Λισαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον χώρο της νόμιμη μετανάστευσης. Το νέο αυτό πλαίσιο μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε σε σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια αυξημένη σημασία της συναπόφασης στον τομέα αυτό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ως νέα Προεδρία του Συμβουλίου θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια επαρκή ε, ένα επαρκή συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μέσω τη Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Η Ευρώπη θέλει να δημιουργήσει μια πολιτική μετανάστευση η οποία είναι ευέλικτη, η οποία θα ανταποκρίνεται στι ανάγκε των αγορών εργασία. Συγχρόνω, ζητώντα να αυξηθεί και η ισότητα ευκαιριών και η κοινωνική συνοχή. Έχει εγκριθεί ήδη το πολιτέ πρόγραμμα, το πρόγραμμα τη Στοχόλμη, για το διάστημα μέχρι το 2014, όπου σαφής στόχος είναι η ανάπτυξη μιας γενικής πολιτικής η οποία βασίζεται στην στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω και να ευχαριστήσω το έργο της Σουηδικής Προεδρίας κατά τη διάρκεια του προηγουμένου εξαμήνου. Ο τρόπος με τον οποίο έχει εκπονηθεί το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι υποδειγματικό σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνειά του θα ήθελα να σας τονίσω ότι το Συμβούλιο αναμένει από την Κομισιόν να παρουσιάσει σε αυτό το εξάμεινο μια ανακοίνωση για το σχέδιο δράσης, η οποία θα υλοποιεί τις βασικές προτεραιότητε αυτού του προγράμματος και θα διατυπώνει σαφείς δράσεις με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και την εφαρμογή του. Τον. Επιτρέψτε μου να σας, εξηγήσω ποιοι είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει στον εαυτό μας ως εξαμηνιαία Προεδρία. Σε συνεργασία με τους Βέλγους και Ούγγρους συναδέλφους μας, η τρόικα λοιπόν αυτών των τριών προεδριών έχουν θεσπίσει δύο βασικούς στόχους των τριών αυτών προεδριών στον τομέα των δικαστικών και εσωτερικών. Πρώτα απ' όλα, να επαναεκκινήσουν οι εργασίες για την νόμιμη μετανάστευση. Δεύτερον, να τεθεί σε κίνηση μια νέα πολιτική ευρωπαϊκή για τα θέματα μετανάστευση. Ένα από τα πρώτα μα καθήκοντα είναι να οργανώσουμε μια πρώτη ετήσια συζήτηση για τι πολιτικέ ασύλου και μετανάστευση για να υπάρχει υποπτία τη εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευση και Ασύλου τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Γι' αυτό βασιζόμαστε στην υποστήριξη τη Κομισιόν και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να αναλύσουμε τι κύριε προόδους που θα επιτευχθούν σε σχέση με αυτό το σύμφωνο η συμβολή της Επιτροπής σας σε, αυτή την άσκηση αξιολόγησης, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι καλόδεκτες. Η έγκριση του σχεδίου για τους ε, ανήλικου, τους μη συνοδευομένους ανήλικους από τρίτες χώρες είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας. Αυτοί οι ανήλικοι που έρχονται από τρίτες χώρες είναι μια ιδιαίτερα τρωτή ομάδα του πληθυσμού η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματά τους. Είναι μια πρόκληση η οποία οδηγεί σε ανησυχίες και απαιτεί μια απάντηση σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να συνδυάζει την πρόληψη, την προστασία και τη βοήθεια για την για τον επαναπατρισμό των ατόμων αυτών, πάντα με γνώμονα το καλύτερο συμφέρον αυτών των ανηλίκων ατόμων. Το Συμβούλιο έδωσε στην Κομισιόν μια σαφή εντολή για την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου, το οποίο θα συμπληρώσει τα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε ήδη. Είμαστε σε επαφή με την γραμματεία της Επιτροπής σα, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, για να εξασφαλίσουμε μια κατάλληλη παρουσία της Επιτροπής σα για ένα θέμα το οποίο έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια. Σε ό,τι αφορά την πτυχή της ενσωμάτωσης, η συνδίκη της Λισαβόνας μας δίνει μια ενισχυμένη νομική βάση για τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίνει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να θεσπίσουν μέτρα ώστε να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη στην προώθηση της ενσωμάτωσης των πολιτών τρίτων χωρών που διαβιούν νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση εφαρμογή της νέας αυτής ευρωπαϊκής πολιτικής ενσωμάτωσης είναι εξάλλου ένας από τους στόχους που έχει θέσει τον εαυτό της η Ισπανική Προεδρία. Για το λόγο αυτό, στις 15 και 16 Απριλίου στη Θαραγώσα θα γίνει η τέταρτη Υπουργική Σύνοδος των Υπουργών Ενσωμάτωσης, όπου θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, ενσωμάτωσης σαν μοχλού κοινωνικής ανάπτυξης και ε, οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη σε εδώ και τη νέα νομική βάση που μα δίνει η Συνδίκη τη Λισαβόνα, καθώ και τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Η δήλωση η οποία προέκυψε από την διάσκεψη η οποία θα προκύψει μάλλον από αυτή τη διάσκεψη, θα τεθεί για επίσημη έγκριση στο Συμβούλιο υπό τη μορφή συμπεράσματων. Τέλος, η Ισπανική Προεδρία θέλει να συνεχίσει τις προσπάθειες στην ανάπτυξη ενός πολιτικού πλαισίου που νόμιμης μετανάστευσης που βέβαια καθυστέρησε αυτή η διαδικασία λόγω της οικονομικής συγκυρίας τους τελευταίους μήνες, αλλά η Ισπανική Προεδρία θα κάνει κάθε προσπάθεια να προωθήσει και πάλι αυτό το θέμα. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν μεγάλη ε, έμφαση στην ε, ρύθμιση της ενιαίας άδεια διαμονής. Πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή της ε, Λισαβόνας είναι θετικό το πλαίσιο για την δημιουργία αυτής της, αυτού του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο απαιτεί και την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το οποίο εξασφαλίζει μια ισόρροπη και ισοδίκια μεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύει λοιπόν η Προεδρία ότι τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν με μεγάλη ταχύτητα να συμφωνήσουν για αυτήν την τόσο σημαντική οδηγία. Η, Ισπανική Προεδρία προφανώς θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Περιμένουμε επίσης ότι και η <clears throat> Επιτροπή σας θα αντιμετωπίσει τις δύο οδηγίες για την νόμιμη μετανάστευση. Καταρχήν για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν αποσπαστεί μέσα στην ίδια επιχείρηση και δεύτερον για τις συνθήκες πρόσβασης και εγκατάστασης ε, πολιτών τρίτων χωρών για μια συγκεκριμένη κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ελπίζουμε ότι και οι δύο αυτές προτάσεις οδηγίες που έχουν παρουσιαστεί από την ε, Κομισιόν θα διεκπαιδευτούν με ταχύτητα, Εμεί θα πράξουμε τα απαραίτητα μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, αυτή είναι και η τομή προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την Ισπανική Προεδρία για την νόμιμη μετανάστευση και την ενσωμάτωση των μεταναστών. Έχουμε ενώπιόν μα σημαντικά καθήκοντα και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι θα κάνω όλα τα απαραίτητα για να υπάρξει μια ρευστή και διάφανη διαδικασία Συνεργασία μαζί σας. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι προφανώς στη διάθεσή σα για να απαντήσω τα ερωτήματα τα οποία τυχόν θέλετε θέση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Προχωρούμε τώρα στον πρώτο γύρο ερωτημάτων. Μία ερώτηση για κάθε πολιτική ομάδα που εκπροσωπείται στην Επιτροπή μας. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης 2 λεπτά το μέγιστο μετά από αυτό το πρώτο χρόνο ερωτήσεων όπου θα λάβει το λόγο ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδα, δεν ξέρω αν θα αυτός θα συντονιστεί ή όχι. Θα απαντήσει ο κύριος υπουργό από κύριους στον πρώτο γύρο και θα περάσουμε μετά σε μεταγενέστερους γύρους ερωτήσεων. Ο Σάιμον Μπουσούτη έχει το λόγο. Uh, thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στην ε, εφαρμογή της ε, Συμφωνίας για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Εμείς όμως θα σας κρίνουμε κύριε Υπουργέ βάσει των δράσεών σας, των πράξεών σας, ε, στο τέλος της Προεδρίας δηλαδή. Και το λέω αυτό γιατί κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενός ενάμιση χρόνου, από τότε δηλαδή που το σύμφωνο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, ελάχιστα απτά πράγματα έχουν γίνει, ελάχιστα αποτελέσματα είδαμε. Εκτός και αν κάνω λάθος, νομίζω ότι ε, μία μόνο νομοθετική πρόταση, του να δημιουργηθεί δηλαδή υπηρεσία ασύλου, μόνο αυτή εγκρίθηκε το παρελθόν έτος. Δεν είναι πολύ καλό αυτό και γι' αυτό σας λέω ότι εμείς θα σας κρίνουμε βάσει απτών αποτελεσμάτων. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε ιδιαίτερα αποτελεσματικός και να λάβετε το ζήτημα αυτό πολύ σοβαρά υπόψη σας. Δύο συγκεκριμένα ζητήματα μας αφορούν κυρίω. Στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασύλου, το ένα έχει να κάνει με την αλληλεγγύη. Η κοινή αυτή πολιτική θα πρέπει να βασιστεί στην αλληλεγγύη. Σήμερα αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα, για παράδειγμα με την πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνου 2, το οποίο έχει μπλοκάρει ουσιαστικά στο Συμβούλιο για παραπάνω από ένα χρόνο. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε για να προχωρήσουμε με την νομοθετική πρόταση. Και βέβαια, το ίδιο το νομοθετικό πακέτο για το άσυλο έχει φτάσει σε ένα διέξοδο και θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Τώρα όσον αφορά το ΕΛΚ περισσότερο, θεωρούμε ότι υπάρχει μια κατάχρηση της πολιτικής ασύλου στη χώρα που ξέρω εγώ καλύτερα. Περίπου 90% των μεταναστών που φτάνουν στην Μάλτα κάνουν αίτηση για άσυλο και είναι σαφές ότι δεν πρέπει να δοθεί σε όλους αυτούς άσυλο. Ελάχιστοι ουσιαστικά καταφέρνουν να έχουν το καθεστώ του πρόσφυγα στο τέλο. Τι πρόκειται να κάνει λοιπόν η Ισπανική Προεδρία για το φαινόμενο αυτό τη κατάχρηση τη κοινή πολιτική ασύλου. Είναι ένα ακόμα ερώτημα που σα θέτω. Κυρία Ρομέρο. Χάμπρικη θα λάβει τη θέση μου. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και κάποιους μήνες ή μάλλον εδώ και κάποια χρόνια, αναφερόμαστε στη δημογραφική προοπτική της Ευρώπης ότι θα χρειαστεί περίπου 50 εκατομμύρια μεταναστών στα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στον κύριο Υπουργό αν η Ευρώπη έχει θέσει το ερώτημα της διοργάνωσης της αντιμετώπισης αυτού του δημογραφικού και πολιτικού και οικονομικού και κοινωνικού επίσης προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα από τα συμπεράσματα τα οποία, στα οποία κατέληξε η ομάδα των σοφών, οι οποίοι εργάζονται πάνω στο θέμα των δημογραφικών προοπτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει το γεγονός ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σχεδιάσει την ενσωμάτωση σε μεγάλο βαθμό μεταναστών τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι όμως αν έχουμε κάποια σχέδια για αυτή την πολιτική ή όχι. Και δεύτερον θέλω να το θέσω αυτό και σε σχέση με το εξής θέμα, κύριε Υπουργέ, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε ορισμένε χώρε, δηλαδή η επιλογή προσοντούχων μονάχα μεταναστών. Αυτή είναι πια μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαγράφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποια σχέδια για την υλοποίηση ή όχι αυτών των ιδεών. Γιατί είναι γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για την μετανάστευση οι οποίες μπορούν να μας προσφέρουν άτομα με δεξιότητες οι οποίες είναι χρήσιμες με την Ευρώπη. Θα ήθελα να ξέρω αν η Ισπανική Προεδρία έχει κάποιες προτάσεις σχέση με τα θέματα αυτά για τους επερχόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Κύριε Λάτφορντ. Θέλετε το λόγο για τους φιλελεύθερους, κύριε Λάτφορντ. Βίξτρομ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας και ιδιαίτερα την δική σας παρουσίαση. Ένας από τους στόχους σας είναι να ενδυναμώσετε την κοινωνική διάσταση, είπατε. Στα πλαίσια της οικονομικής λοιπόν κρίσης, όντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους και Καταλαβαίνετε ότι υποστηρίζοντα του ανθρώπου αυτού θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε και την κοινωνική διάσταση, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε στα πλαίσια τη μετανάστευση και του ασύλου και να αντιμετωπίσουμε τι σχετικέ προκλήσει. Επομένω, θα ήθελα να γνωρίζω ποια διασύνδεση βλέπετε ανάμεσα στην μετανάστευση, την ενσωμάτωση και μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Thank you. Señor Romeva, por los verdes. Muchas gracias. Muy brevemente, tres. Ευχαριστώ. Με μεγάλη ταχύτητα τρει ή τέσσερι ερωτήσει πάρα πολύ συνοπτικά και σύντομα. Καταρχήν, δεν αναφερθήκατε στο θέμα αυτό, θα ήθελα να μα πείτε τι προβλέπετε για συγκεκριμένα μέτρα όπως χάρη η πρόσληψη στην χώρα προέλευση των μεταναστών. Δεύτερον, Αναφερθήκατε στο θέμα τη οικογένειακή επανένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε καιρού κρίση και εκεί αυτέ οι οικογένειε πλήττονται ιδιαίτερα λόγω τη δυσκολίες που έχουν αυτά τα άτομα για να μπορέσουν να επιτύχουν κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ότι είναι ένα δικαίωμα η επανένωση των οικογενειών. Τρίτο ερώτημα, πάλι πολύ συγκεκριμένο, ένα από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν την ομάδα μας είναι η κατάσταση στα κέντρα κράτησης. Σε ορισμένες χώρες η κατάσταση είναι ικτρή <clears throat> και βλέπουμε να υπάρχει και σημαντική επιδείνωση στην περίπτωση πολλών χωρών και ένα νομικό λίμπο, γιατί η κατάσταση κράτησης δεν είναι ούτε νόμιμη ούτε παράνομη. Και επομένως το ερώτημα είναι αν υπάρχει μια προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα κέντρα κράτης. Μια τελευταία ερώτηση πιο πολιτική. Είδαμε μια πρόταση να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο ένα είδος αντιμετώπισης των Δήμων, από την πλευρά των Δήμων, των ατόμων οι οποίοι δεν έχουν νόμιμες συνθήκες ε, διαβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα το αντιμετωπίσει συνολικά αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σταβάρες, κύριε Υπουργέ. Καλό απόγευμα κύριε Υπουργέ Σάβης, Τσάβες μάλλον. <clears throat> Είδαμε γεγονότα στο Ροζάνο, στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια των εορτών. Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε. Ένα είδος καταδίωξης των μεταναστών ή είτε ε, νομίμων είτε παρανόμων που έχασαν την εργασία τους εποχιακού χαρακτήρα. Εδώ θα ήθελα να ξέρω συγκεκριμένα τι αναμένει ο κύριος υπουργό από την οδηγία που προαναφέρατε συγχρόνως. Αν τα προβλήματα αυτό που είδαμε στο Προζάνο επαναληφθούν και σε άλλες χώρες, είναι δυνατόν με πολιτικές περιοριστικές περιορισμού της μετανάστευσης σε μερή ρεαλιστικές πολιτικές μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ή θα καταλήξουμε να δημιουργήσουμε τεράστια γκέτο παράνομων μεταναστών τα, οι οποίοι θα είναι στο έλεος των εκμεταλλευτών εργοδοτών τους. Επίσης, αναφερθήκατε και στο θέμα της, μετανα... της των μεταναστών και αυτό είναι πράγματι ένα από τα βασικά στοιχεία μιας δημοκρατία, όπως ξεκινάει και από την Αμερικανική Επανάσταση, no taxation without representation, όποιος ζει σε μια χώρα και πληρώνει φόρους, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα του εκλέγην και του Θα Αναφέρομαι στους νόμους μετανάστες, οι οποίοι συμβάλλουν με τους φόρους τους στην κοινωνική ζωή μιας χώρας, δεν θα πρέπει αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα κοινά στη χώρα όπου ζουν. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την παράνομη μετανάστευση. Η μαζική νομιμοποίηση των μεταναστών λαμβάνει χώρα σε διάφορα κράτη-μέλη. Πριν από λίγα χρόνια, στην Ισπανία, νομιμοποιήθηκαν χιλιάδες μετανάστες και άλλες χώρες ε, προβαίνουν σε αντίστοιχα μέτρα. Αυτό το πρόβλημα ε, δεν ενθαρρύνει τη λαθρομετανάστευση. Και τότε αυτό το πρόβλημα περνάει από το ένα κράτος στο άλλο, στο άλλο κράτος μέλος. Μέσω της ελεύθερης μετακίνησης δηλαδή, αυτοί οι λαθρομετανάστες περνάνε από το ένα κράτος στο άλλο κράτος μέλος και το πρόβλημα ε, μεταβιβάζεται τροποντινά στην άλλη χώρα. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ε, έγκυρης προειδοποίησης τουλάχιστον για να ενημερωθεί το άλλο κράτος μέλος ότι πρόκειται να υπάρξει αυτή η κίνηση. Νομίζω ότι υπάρχουν ελλείψεις στο σύστημα. Γιατί δεν υπάρχει συνένεση α, της μίας χώρας ε, στην διαδικασία νομιμοποίησης της διπλανής χώρας, της όμορης χώρας. Η Ισπανική Προεδρία σκοπεύει να κάνει κάτι για αυτό το πρόβλημα. Ωραία. Ένας πρώτος γύρος απαντήσεων, κύριε Υπουργέ. Έχετε ακούσει ένα εκπρόσωπο από κάθε πολιτική οικογένεια και έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι στο τέλος της Ισπανικής Προεδρίας, στο τέλος του εξαμήνου μας και όταν θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Θα πρέπει να επανέλθω ενώπιον σας και να αναφερθούμε στα θέματα αυτά. Είναι σαφές ότι το θέμα της, ε, του συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει ότι για πρώτη φορά όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση που έχει την υποστήριξη της πολιτικής θέλησής μας. Χρειάζεται όμως να διατρέξουμε αρκετό δρόμο και θα πρέπει να αναπτύξουμε τα στοιχεία αυτού του πακέτου και να δούμε ποια θα είναι η αξιολόγηση της Κομισιόν για ό,τι αφορά στο θέμα της παροχής ασύλου, εμείς ως Προεδρία τονίσουμε ότι θέλουμε μια τακτική και νόμιμη μετανάστευση. Και επομένως, αν η μετανάστευση είναι οικονομική, συνδέεται με την εργασιακή αγορά αν πρόκειται για αίτηση ασύλου, θα πρέπει να συντρέχουν οι συνθήκες που αιτιολογούν αυτό το άσυλο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κατάχρηση της αίτηση ασύλου. Αυτή είναι λοιπόν η οπτική γωνία της Ισπανικής Προεδρίας, ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί περισσότερους μετανάστες σε ένα ε, προσεχές μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια προβληματική για τα θέματα αυτά. Δεν είναι σωστό να βλέπουμε τη μετανάστευση μονάχα μέσα σε ένα συγκυριακό πλαίσιο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή με την οικονομική κρίση έχει μειώσει σημαντικά τις προσδοκίες που είχε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Λισαβόνας. Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κρίση, είναι πάνω από 8 εκατομμύρια ατόμων που έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους. Αυτό Σημαίνει ότι αν έχουμε 8 εκατομμύρια ανέργους, θα πούνε κάποιοι γιατί να σκεφτούμε για τη μελλοντική μετανάστευση. Είναι σίγουρο όμως ότι σε ένα βραχυπρόθεσμο επίπεδο ο στόχος μας θα πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τη θέση εργασία τους, είτε είναι Ευρωπαίοι είτε μετανάστες, να ξαναβρούν θέσεις εργασίας. Σε σχέση όμω με ένα πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει την οικονομική τη ανάπτυξη και για να γίνει κάτι τέτοιο θα είναι απαραίτητο να υποδεχθεί και μετανάστε, άτομα τα οποία θα μοιραστούν <clears throat> τη ζωή στι χώρε μα και θα εργαστούν εδώ. Για τη μετανάστευση ατόμων με ειδικά προσόντα. Είναι σημαντικό αυτό. Αλλά βρισκόμαστε σε ένα κοινοβουλευτικό χώρο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα ήταν σωστό από την πλευρά της Ευρώπης να να ζητούμε από τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν αποδώσει κάποιους πόρους για να εκπαιδεύσουν ορισμένα μέλη του πληθυσμού τους, κυρίως το υγειονομικό προσωπικό, ενώ αυτές οι χώρες έχουν κάνει αυτές τις προσπάθειες να εκπαιδεύσουν αυτό το προσωπικό, εμείς τους προσελκύσουμε στην Ευρώπη για να διατηρήσουμε το κράτος ευμάριάς μας, με τον τρόπο αυτό κατακριμνίζοντας τις συνθήκες ευμάρειας στις χώρες προέλευσης. Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια ροή, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε υπόψη μας, να έχουμε υπόψη μας και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα προέλευσης. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα τα οποία τέθη σε σχέση με τη λεγόμενη μπλε κάρτα και αφορούσε το υγειονομικό προσωπικό. Να υπάρξει και μία ανάλυση των συνδικών στη χώρα προέλευση, η ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή και η ενσωμάτωση των μεταναστών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ευρώπη είναι ένα χώρο κοινωνικό μέσα στον οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα και σε περίπτωση κρίσης οικονομικής να μην τεθεί ένα αμφιβόλο η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας χώρος κοινό τον οποίο εμείς θα πρέπει να τον συμμεριζόμαστε με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Από τη στιγμή όμως που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να εξασφαλίσει ότι θα γίνει πράγματι αυτή η ενσωμάτωσή τους, ώστε τα άτομα αυτά να μην απαρνηθούν την ταυτότητά τους, αλλά ούτε να υπάρξουν συγκρούσεις σε επίπεδο καθημερινής διαβίωσης. Αυτή είναι η πιο σημαντική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η διαχείριση του φαινόμενου της μετανάστευσης. Γιατί πρέπει να υπάρξει ευκυβερνησία στο, στη μετανάστευση. Πρόσληψη εργαζομένων ήδη στη χώρα προέλευσής τους. Αυτή είναι ίσως η καλύτερη λύση για να υπάρξει τακτικός χαρακτήρας στη μετανάστευση. Προσλαμβάνουμε κάποιον που βρίσκεται ακόμα στη χώρα του και όταν τελειώσει η περίοδος για την οποία έχει γίνει η πρόσληψη αυτού του ανθρώπου, είναι δεσμευμένος να επανέλθει στην χώρα του. Μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα της ε, Ισπανίας. Κάθε χρόνο προσλαμβάνουμε 30.000 άτομα στο Μαρόκο για να εργαστούν σε γεωργικές εργασίες. Και τα άτομα αυτά επανέρχονται στο Μαρόκο όταν τελειώσει αυτή η καλλιεργητική περίοδος. Η περίοδος μάλλον στην Ανταλουσία. Επομένως αυτό είναι ένα παράδειγμα για το θέμα της ε, πρόσληψης στη χώρα το θέμα της οικογενειακής επανένωσης είναι κάτι το οποίο ποικίλει βέβαια από χώρα σε χώρα, αλλά υπάρχει ένα κοινό, ένας κοινός που πρέπει να το λάβουμε υπόψη, δηλαδή να υπάρξει ενίσχυση της επανένωση του οικογενειακού πυρήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα άτομο να μπορεί το ταχύτερο δυνατό να ζει μαζί με τον πυρήνα της οικογένειάς του, δηλαδή με την σύζυγό του ή τον σύζυγό του και τα παιδιά του. Και τώρα η ενσωμάτωση, η επανένωση και των γονέων και της ευρύτερης οικογένειας, αυτό είναι ένα άλλο πιο ευρύ θέμα. Εμεί κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του πυρήνα της οικογένειας, της πυρηνικής οικογένειας όπως λέγεται και της επεκτεταμένης οικογένειας. Για τα κέντρα κράτησης, <clears throat> είναι περισσότερο στην αρμοδιότητα του συναδέλφου μου, αλλά σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητά μας εμείς προσπαθούμε, όπως είναι σαφές, να έχουν αυτά τα κέντρα κράτησης ένα χαρακτήρα όχι σοφρονιστικού καταστήματος, αλλά ενός χώρου όπου μπορούν να είναι σεβαστές οι αρχές της νόμιμης μετανάστευσης, του, ότι είναι νόμιμη μετανάστευση. Τώρα για την περίπτωση του ΒΙΚ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αρνηθεί ένας Δήμος να καταγράφεται στα μητρώα του Δήμου ένα άτομο ανεξάρτητα από το νομικό του καθεστώς. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξουν καταχρήσεις αρμοδιοτήτων στην περίπτωση αυτή. Για τους εποχιακούς εργαζομένους τέλος, η Προεδρία αναμένει από την Κομισιόν να παρουσιάσει ένα έγγραφο, ένα σχέδιο οδηγίας το οποίο θα ρυθμίσει το θέμα των εποχιακών εργαζομένων. Αποδίδουμε μια τεράστια σημασία στο θέμα αυτό γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να τύχει ρύθμιση ώστε αυτός ο εποχιακός χαρακτήρας ή ο προσωρινός χαρακτήρας να μην οδηγήσει σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Και σε σχέση με το δικαίωμα του εκλέγην, θα σας πω ότι είναι αυτό το οποίο εγώ υποστήριξα σαν δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Καταλωνία και στη συνέχεια σαν υπουργό. Υποστηρίζω στις δημοτικές εκλογές να ψηφίζουν οι μετανάστες. Νομίζω ότι αν δεν αναγνωρίζετε αυτό το δικαίωμα, απομακρύνουμε το μετανάστη από την πραγματικότητα μέσα στην οποία διαβεί. Και φυσικά από εκεί και πέρα εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει την νομοθεσία του και τις συγκεκριμένες ρήτρε για τα θέματα αυτά. Τέλος. Η συμφωνία μας δεν επιτρέπει την μαζική ρύθμιση για τους μετανάστες. Λέει ότι τα κράτη-μέλη τα οποία υπογράφουν αυτή τη συμφωνία δεσμεύονται να μην προχωρούν σε μαζικές νομιμοποίησεις μεταναστών. Σε κάποιες στιγμές οικονομικής ανάπτυξης στο παρελθόν είχαν γίνει τέτοιες μαζικές νομιμοποίησεις για να ομαλοποιηθούν οι καταστάσεις ομάδων ατόμων. <clears throat> Νομίζω όμως αυτή τη στιγμή η Ευρώπη εν ώψη του μέλλοντος θα πρέπει να προχωρήσει στην ρύθμιση μιας νόμιμης, ελεγχόμενης και τακτικής μετανάστευσης και πάντα με ένα συμβόλαιο εργασία στην χώρα προέλευση. Νομίζω ότι αυτέ είναι οι βασικέ σκέψει που υπήρχαν πίσω από την εκπόνηση του συμφώνου και εμεί πρέπει να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Προτείνω να προχωρήσουμε όπω κάναμε και προηγουμένω, με τον Υπουργό Εσωτερικών, να έχουμε ένα δεύτερο γύρο όπου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε δυνατότητα να μιλήσουμε ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμό μελών της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών που ζήτησαν το, το λόγο και θα ακολουθήσει μια ομαδική απάντηση στα ερωτήματά τους από την πλευρά του κυρίου Υπουργού. Προτείνω λοιπόν πρακτικά για να καλύψουμε το μεγαλύτερο αριθμό ερωτώντων να υπάρχει χρόνος ερώτησης ενός λεπτού και μόνο. Ο κύριος Δίας Δεμέρα καταρχήν. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ και καλή τύχη στα εγχείρημά σας. Όλοι οι μετανάστες, οι παράνομοι, οι λαθρομετανάστες έχουν κοινωνικές ανάγκες, όλοι τους. Έχουν το δικαίωμα με κεφαλαία να τις καλύψουν σε ορισμένα καθημέλια, ενώ σε άλλα όχι. Η ενσωμάτωσή τους που είναι μέσα στις αρμοδιότητές τους. Η ενσωμάτωση στην οποία αναφερθήκατε περιλαμβάνει την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών τους, των ζωτικών τους αναγκών ή σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων ή αυτό αφορά μονάχα τους ε, νόμιμους μετανάστες. Για να υπάρχει μια κοινή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ρυθμίσουμε ένα νόμιμο χώρο εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πώς είναι αυτοί και ποιοι είναι αυτοί που θα είναι νόμοι. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα στις τρεις ε, πρόεδρες της Τρόικας. Λάτσεβιτ Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που μιλήσατε πολύ συγκεκριμένα για τις προτεραιότητες για την μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών. Με μεγάλη χαρά άκουσα τις υποσχέσεις σας για τους επόμενους έξι μήνες της Προεδρίας σας. Δηλαδή, θα εξασφαλίσετε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν θα πρέπει να... Δεν θα χρειάζεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα προβλήματα θα επιληθούν. Θα ήθελα επίση να με καθησυχάσετε ότι θα λάβετε πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την οδηγία του Συμβουλίου για την πρόταση να εκδοθεί μία άδεια σε υπηκόους των χωρών για να διαβιούν και να εργαστούν ε, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα υπάρχει μία διαδικασία ε, για αυτούς τους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της ε, Γαλλικής Προεδρίας έγιναν κάποιοι συμβιβασμοί, αλλά κατά τη διάρκεια της Τσεχικής και Σουηδικής Προεδρίας δεν έγινε τίποτα για αυτό το θέμα. Έχετε κάποια μυστικά όπλα, κάποιους μυστικούς άσους, Πρόεδρε, ε, κύριε Υπουργέ, ούτω ώστε να φτάσουμε σε συμβασμό μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και να υιοθετηθεί τελικά αυτή η οδηγία κατά τη διάρκεια τη προεδρία σα. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τι εξήγησει που μα δώσατε. Εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω μετά την έγκριση της συνθήκη Λισαβόνα, πώ θα αντιμετωπιστεί στην σχεδιοποίηση των πολιτικών μετανάστευση, πώ θα αντιμετωπιστεί το θέμα των διοικητικών αρχών οι οποίες βάσει της αρχής της επικουρικότητας είναι αυτές αρμόδιες να δώσουν τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα αυτά τα οποία ζουν στην Ευρώπη. Επομένω, τα κράτη καθορίζουν την πολιτική μετανάστευσης, αλλά οι πιο κοντά στον πολίτη υπηρεσίες, οι περιφερειακές ή οι τοπικές, θα δώσουν τις υπηρεσίες στον μετανάστη. Πώς θα γίνει αυτό μέσα στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας. Δεύτερον, αναφέρατε την ανάγκη που έχουμε για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης ...την παρουσία των μεταναστών. Μήπως θα πρέπει να αναπτύξουμε και μια καμπάνια συνειδητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών για να αποφύγουμε την δημαγωγική εκμετάλλευση του φαινομένου της μετανάστευσης, κάτι που γίνεται πολύ συχνά. Και τέλος, η ενσωμάτωση των ανηλίκων στα κέντρα για τους ε, ανηλίκους. Υπάρχουν κέντρα κατάρτισης, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ότι τα κέντρα που δίνουν την καλύτερη κατάρτιση έχουν τόσους μετανάστες ανήλικους που δεν μπορούν να δώσουν σοβαρή κατάρτιση. Υποστηρίζετε να υπάρχουν ποσοστό σε ανακράτο για αναπεριοχή για να υπάρχουν καλύτερε υπηρεσίε, οι οποίε δίνουν στου μετανάστες. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ποιε είναι οι προτάσει σα πολύ συγκεκριμένα τι θα κάνετε ούτως ώστε τα κράτη-μέλη και η, το, η Frontex να μην προωθήσουν τα μέτρα επαναπρόθεσης ε, στα σύνορά μας. Ε, την περασμένη άνοιξη υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η Frontex προέβησε επαναπροωθήσεις. Θα το διερευνήσετε. Και αν τα κράτη-μέλη ε, δεν ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες για την επαναπρόθεση, τι θα κάνετε, ε, καθώς και για τα συστήματα Ε, Κύριος Γιακολίνου, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να αναγνωρίσουμε την ε, σχέση και συνάφεια ανάμεσα στην παρέμβαση που έκανε ο Υπουργό ε, Ένταξης και ο Υπουργό Εσωτερικών. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων και στενή συνεργασία βεβαίως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, στην Ιταλία υπάρχουν πέντε ε, εκατομμύρια ε, λαθρομεταναστών που έχουν ε, νομιμοποιηθεί. Και επίσης 250.000 ε, επιχειρήσεις ε, προσλαμβάνουν τέτοιους ε, λαθρομετανάστες. Θα σταματήσουμε. Τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Επίσης, το έγγραφο για τη Στοκχόλμη Μιλάει για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και για την ίση κατανομή των μεταναστευτικών ροών. Ποιε είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ τη Ισπανική Προεδρία για αυτό το θέμα. Δεν ξεχνάω την όλο και αυξανόμενη κοινωνική προστασία των μεταναστών που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ναγκόμες. Δεν είναι εδώ. Signora Kinga Κυρία Κίνγκα Γκάντς. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αυτές οι τρεις προεδρίες και η Ισπανία, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα της ε, μετανάστευσης και ασύλου. Πώς θα προχωρήσουν. Εσείς είστε η πρώτη προεδρία από την ε, Τρόικα που αναφέρατε. Πώς θα υλοποιήσετε αυτή την πολιτική. Πώς μπορείτε να προωθήσετε τις προτεραιότητε που αναφέρθηκε ότι είναι οι προτεραιότητε τη Ισπανική Προεδρία. Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα τι εφαρμόσετε. Κυρία Φλότχο, ε, είσαστε υπεύθυνο για την απασχόληση και τη μετανάστευση. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η χω, ο συνδυασμό αυτό. Ε, το συζητάμε και στη χώρα μου. Μετανάστευση και εθνική ταυτότητα. Λοιπόν, στην Ευρώπη, ξέρετε, ε, αναφερθήκατε στα 30.000 άτομα που έρχονται στην Ανδαλουσία για να μαζέψουν τις φράουλες. Νομίζω ότι οι μετανάστες στην Ευρώπη ε, θέτουν διάφορα ερωτήματα. Έχουμε λαθρομετανάστες που όμως έχουν ε, νόμιμες ε, άδειες εργασίες που πληρώνουν ε, φόρους και εισφορές. Θα πάρετε μια πρωτοβουλία ούτως ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι μετανάστες στην Ευρώπη να διαμένουν νομίμως γιατί ακριβώς έχουν έμιστη εργασία η οποία είναι απόλυτα νόμιμη. Έπειτα, μια άλλη κατάσταση είναι η κατάσταση του Ροζάρνου. Εκεί το 80% ε, είναι νόμιμοι μετανάστες ε, που διαμένουν νόμιμα στην Ευρώπη αλλά που δουλεύουν ε, μέσα σε συνθήκες δουλείας, χωρίς καμία σύμβαση εργασίας. Θα πάρετε λοιπόν μια πρωτοβουλία ούτως ώστε αυτά τα άτομα τα οποία βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη να τακτοποιηθούν σε ό,τι αφορά την εργασία τους, των συνθήκων εργασίας τους, να διαμένουν νόμιμα στην Ευρώπη. Τι θα κάνετε για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για την οικονομική μετανάστευση. Λες και είναι ε, ευγενής μετανάστευση και αλτρουιστική. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Οι τοπικοί καπιταλιστές εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους σαν να είναι μέσα παραγωγής και όχι άνθρωποι. Ε, στα, αποσταθεροποιεί τις χώρες ε, υποδοχής, ε, δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά εργασίας, ε, μειώνει τους μισθούς. Και επίσης δεν τους δίνει τις απαραίτητες δεξιότητες. Δεν νομίζω ότι είναι η προτιμητέα λύση της διακίνησης ανθρωπίνων όντων. Στην πραγματικότητα είναι μια μορφή αυτής της παράνομης διακίνησης ανθρωπίνων όντων. Κυρία Ναγκόμες, προηγουμένως σας δώσω το λόγο, δεν ήσασταν εδώ. Ε, θα σας δώσω τέλος πάντων τώρα την ευκαιρία να μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω μέσα στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας αν έχετε τον στόχο να προωθήσετε την νόμιμη ενσωμάτωση των μεταναστών. Εμείς στην Πορτογαλία έχουμε και σε άλλες χώρες άτομα που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το καθεστώς τους. Είναι τα άτομα τα οποία δεχτήκαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Γουαντάναμο. Και είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα εκπροσώπους από την Αμερικανική κυβέρνηση οι οποίοι συζήτησαν μαζί μας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξέρω. Βέβαια αφορά μονάχα έξι ευρωπαϊκές χώρες που υποδέχτηκαν κρατούμενους από το Γουαντάναμο, μία από τις οποίες είναι η Ισπανία. Με τι καθεστώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει δεκτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτικοί πρόσφυγες, ως μετανάστες και μέσα στη νέα βάση τη νομική της συνθήκης της Λισαβόνας. η οποία θέλει να υπάρξει πρόθεση της ενσωμάτωσης των ατόμων αυτών έχει κάποια αμνία για μια πολιτική, όχι ατομική, αλλά μια πολιτική σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Για μια κοινή απάντηση. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό σε όλα αυτά τα διάφορα θέματα τα οποία ετέθησαν από τους προλαλήσαντες. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Το θέμα της ενσωμάτωσης και των κοινωνικών αναγκών των μεταναστών είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα από την πλευρά της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη είναι προφανές ότι <clears throat> θα πρέπει να είναι η βάση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου λόγου, παγκόσμιας αντιμετώπισης, όπου οι ιδέες αυτές θα είναι αποδεκτές από όλους και ότι θα ακολουθηθεί αυτή η βέλτιστη πρακτική. Η ολοκλήρωση πρέπει να γίνεται πάντα στο πιο πλησίον επίπεδο προς το μετανάστη. Αλλά πρέπει συγχρόνως να έχουμε και μια πιο συνολική θεώρηση. Το θέμα της εργασιακής αγοράς, νομίζω ότι εδώ η πρώτη μου απάντηση ήταν ότι η μετανάστευση θα πρέπει πάντα να είναι σε σύνδεση με την εργασιακή αγορά με τις εξελίξεις στην αγορά αυτή που προσδιορίζουν και τις ανάγκες που υπάρχουν. Η Ευρώπη <clears throat> θα πρέπει φυσικά να έχει και μια προοπτική, γιατί η Ευρώπη έχει τον στόχο της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής θα πρέπει να έχει ένα οικονομικό μοντέλο, ένα μοντέλο παραγωγής και μια σειρά από στόχους. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν και οι ανάγκες που έχει η Ευρώπη στο εργασιακό επίπεδο και επομένως τις ανάγκες σε μετανάστες εργαζόμενους. Στο θέμα των ανηλίκων. Υπάρχει η αρχή που λέει πάντα ότι πρέπει να αποφύγουμε οι μαφίες να... Πρέπει να αποφύγουμε οι μαφίες να χρησιμοποιούν τους ανήλικους μέσα σε αυτή τη λαθρεμπορία ανθρώπων που συμβαίνει πολλές φορές. Δηλαδή πολλές φορές πίσω από ένα ανήλικο δεν υπάρχει η προσωπική απόφαση αυτού του νέου να προσπαθήσει να βρει μια καλύτερη μοίρα. Πολλές φορές υπάρχει μια μαφία <clears throat> η οποία τον παρακινεί και τον βοηθά ακόμα για να μεταναστεύσει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά δεν μπορούμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε τον ανήλικο ως μετανάστη. Ο ανήλικος είναι πρώτα απ' όλα ανήλικος και επομένως εδώ θα πρέπει να υπερισχύσει αυτή η αρχή της ειδική μεταχείρισης που θα πρέπει να έχει. Και επιπλέον φυσικά θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι τα θέματα των ασυνόδευτων ανηλίκων θα αντιμετωπιστούν πλήρως μέσα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρώπη τα θέματα των ασυνόδευτων ανηλίκων τα έβλεπε στην περίπτωση των χωρών αυτών οι οποίες λόγω της εγκύτητός τους σε ορισμένα σύνορα υφίστανται αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Πρέπει η Ευρώπη να κατανοήσει ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να περιοριστεί μονάχα σε μια χώρα ή σε μια ομάδα χωρών, αλλά θα πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο θα ενδιαφέρει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας και την εσωμάτωση των μεταναστών στην Ευρώπη, εδώ είναι προφανές και τον και από μία ερώτηση ότι πρέπει να υπάρχει <clears throat> μια ποσόστοση αναχώρα, αναπεριοχή για την κατανομή των ανήλικων. Εμείς συζητούμε και θα συζητήσουμε και στη διάσκεψη της Σαραγώσας 3 Μαρτίου για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω στην Ευρώπη διαμορφώνεται όλο και μεγαλύτερη συνένεση ότι <clears throat> το σύνολο των πολιτικών της θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων και επομένως <clears throat> να υπάρξει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος αυτού για την ίδια την Frontex. Εκεί ο στόχος μας είναι ένα στόχο, ο οποίος δεν βρίσκεται στι δικέ μου αρμοδιότητε, Είναι αρμοδιότητα των Υπουργών Εσωτερικών και ο προκάτοχός μου εδώ ενώπιόν σα τα ανέφερε. Αλλά πιστεύω ότι η Ισπανική κυβέρνηση αυτό το οποίο θα προωθήσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της είναι ότι πρέπει να εγκυροποιήσουμε την αρχή της νομιμότητος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διοικητικές ε, αριθμίες κατά κάποιο τρόπο που μπορεί να οδηγήσουν στα άτομα αυτά να κρατούνται, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει νομιμότητα στην δραστηριότητα της Frontex. Εγώ δεν έχω ότι η Frontex δρά με τρόπο απόλυτα νόμιμο και τακτικό. Για το θέμα του Ρωσάρνο που αναφέρθηκε στην, στην Ιταλία, ή μάλλον για το θέμα της ε, νομιμοποίησης. Τίθεται το θέμα του πώς η Ευρώπη θα μπορούσε συνολικά σε επίπεδο θεσμικό οικονομικό να αντιμετωπίσει την απαραίτητη ισορροπία σε ό,τι αφορά την ε, στάση της Ευρώπης για το πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο <clears throat> είναι το καλύτερο εργαλείο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Εδώ έχουν συνενωθεί πολλές πολιτικές αντιμετωπίσεις για τα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητοι οι κανονισμοί και οι οδηγίες, αλλά συγχρόνως πολλές φορές προχωρούμε <clears throat> με το να έχουμε μια κοινή και αλληλέγγυα πολιτική θέληση. Υπήρξε ένα άλλο ερώτημα σχέση με το οποίο πρέπει να σας τονίσω ότι και με το Βέλιο και την Ουγγαρία τις επερχόμενες προεδρίες. Λοιπόν, υπάρχει απόλυτη συμφωνία σε σχέση με τα θέματα αυτά που είναι στην αρμοδιότητά μου. Έχουμε εργαστεί για αυτά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε περιοδικές συναντήσεις με τις χώρες αυτές. Και μπορώ να σας πω ήδη ότι σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μας σε σχέση με τις κατευθυντήρες γραμμές της πολιτικής δράσης της Προεδρίας κατά τη διάρκεια αυτών των 18 μηνών. Και τόσο το Βέλγιο όσο και η Ισπανία έχουμε συλλέξει εμπειρίες και έχουμε γνωρίσει μια εμπειρία σημαντική λόγω του υψηλού επίπεδου ποσοστού μάλλον μεταναστών στις χώρες μας. Για το θέμα των ε, <clears throat> εργαζομένων των συμβάσεων και της διαμονής τους, Αυτά εν μέρει εξαρτώνται και από το Κοινοβούλιο στο βαθμό που θα μπορέσει να προωθήσει το ζήτημα αυτό της ενιαίας άδεια για τους μετανάστες στην πρώτη ανάγνωσή του που θα πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον. Η Ισπανική Προεδρία θα ήθελε να ζητήσει το ταχύτερο δυνατό να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα θέματα αυτά και στη συνέχεια την έγκριση της οδηγίας αυτής η οποία θα επιλύσει τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουν τεθεί. Τέλος, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι η οικονομική μετανάστευση <clears throat> έχει όλα αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα που ανέφερε ο κύριος Βουλευτής. Νομίζω ότι έχει αμφίδρομα θετικά αποτελέσματα και για τη χώρα προέλευσης, διότι επιτρέπει κάποια άτομα να εργαστούν έξω από αυτή τη χώρα και να επανέλθουν έχοντας αποκομίσει μια εμπειρία, μια γνώση και βοηθώντας την οικονομία της χώρας προέλευσης με τα εμβάσματά τους, ενώ συγχρόνως εργαζόμενοι συμβάλλουν στην ευμάρεια της χώρας υποδοχής. Και επίσης, ένα άλλο θέμα που τίθεται, για το Γουαντάναμο αυτό εκφεύγει ολοκληρωτικά των αρμοδιοτήτων μου και γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είναι θέμα ούτε μετανάστευσης ούτε ενσωμάτωσης. είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε στο Συμβούλιο Εσωτερικών, αλλά όχι εγώ προσωπικά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον Υπουργό Ενσωμάτωση και Μετανάστευση, ο οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα αυτά. Τον ευχαριστώ για την παρουσία τη ατζέντα τη Ισπανική Προεδρία για του επόμενου έξι μήνε, για την προσπάθειά του να έχει μια συνθετική σειρά απαντήσεων στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από του βουλευτέ κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασή μα. Έχουμε καθυστερήσει ήδη μισή ώρα σε σχέση με το προβλεπόμενο ωράριο. Επομένως, νομίζω ότι ερμηνεύω την θέληση των μελών της Επιτροπής μας. Μπορούμε κλείνοντας τη συζήτηση να ευχαριστήσουμε τον κύριο Υπουργό και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην υλοποίηση αυτής της ατζέντας που μας παρουσίασε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει όπως σας είπα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να επιταχύνουμε για τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε στο σημείο 5. Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πακιστάν. Τον Οκτώβριο πέρυσι το Κοινοβούλιο έλαβε την συμφωνία και έπρεπε να γνωμοδοτήσει. Η συμφωνία υπεγράφει δύο εβδομάδες μετά. Δεν ήταν δυνατό εμείς να γνωμοδοτήσουμε πριν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και έκτοτε περιμένουμε να μας στείλει το Συμβούλιο την επίσημη απόφαση συμφωνίας Ξέρουμε ότι έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου, επομένως είναι υποχρεωτική η δική μας σύμφωνη γνώμη για να συναυθεί η συμφωνία. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 218, παράγραφος 10, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα. Είναι η πρώτη συζήτηση λοιπόν που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και αυτό θα γίνει και με τις υπόλοιπες συμφωνίες επανεισδοχής που βλέπετε στον κατάλογό μας, στον πίνακα αυτό που σας έχει δοθεί. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια στον εκπρόσωπο της Προεδρίας και στη συνέχεια στον εισηγητή μας, τον κύριο Σόγκορ. Ο κύριος Μπουζουτήλ μου λένε μάλλον ότι είναι ο εισηγητής. Είστε εσείς ο συγητής κύριε Μπουζουτήλ. Αντικαθιστάτε τον κύριο Σόγκορ, τον εισηγητή, μάλιστα. Πρώτα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Πίτερ Μπόσκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο για αυτό το θέμα της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πακιστάν. Ε, και ορίζω και τον κύριο Μπουσουτήλ. Δόθηκε εντολή στην Κομισιόν πριν από 10 χρόνια σχεδόν. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να φτάσουμε σε συμφωνία με το Πακιστάν. Ήταν πολύ δύσκολο να φέρουμε το Πακιστάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μετά όμως από έξι επίσημους γύρους το 2007 ε, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα κείμενο, κάτι που δεν είναι καθόλου προφανές. Εν συνεχεία, ε, περάσαμε και σε άλλες φάσεις. Ε, η μονογραφή της συμφωνίας ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά τελικά ε, υπεγράφει η συμφωνία τον Οκτώβριο του 2009. Και τώρα είμαστε στη τελική φάση. Ελπίζουμε για την οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας επανεισδοχής. Μία συμφωνία επανεισδοχής που είναι εξόχως σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πακιστάν είναι μια χώρα όπου ε, από την οποία είτε ορμώνται οι λαθρομετανάστευς ή ε, περνούν μέσα από αυτήν. Υπάρχουν περίπου 13.500 άνθρωπα που συλλαμβάνονται στα 27 κράτη-μέλη και όλα τα κράτη-μέλη θέλουν να εξασφαλίσουν το γρήγορο και αποτελεσματικό, τη, τη γρήγορη και αποτελεσματική επιστροφή. Και αυτό το καταφέραμε σε 4.000 περιπτώσεις. Δεν πρόκειται μόνο για μια συμφωνία επανειστοχής που αφορά τους υπηκόους του Πακιστάν, αλλά όπως θα έχετε δει και σε ένα άρθρο ε, που αφορά ε, την επανεισδοχή υπηκών τρίτων χωρών και απάτριδων, πιστεύουμε ότι είναι ε, γενικά μεγάλο επίτευγμα για τις διαπραγματεύσει νομίζουμε ότι σε αυτή τη, ε, συγγνώμη, σε αυτή τη φάση διαπραγματευόμαστε και μια συμφωνία επανεισδοχή με την Τουρκία. Η Τουρκία επίσης είναι μια άλλη πολύ σημαντική χώρα. Ο Γενικός μας διευθυντή, ο κ. Φόρ, θα πάει στην Άγκυρα, μάλλον στις 19 του Φεβρουαρίου, για να ξαναρχίσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για μια τέτοια συμφωνία επανεισδοχή. Το Πακιστάν για τους Τούρκους ε, συναδέλφους είναι πολύ σημαντική χώρα προέλευσης μεταναστών. Επομένως, το ότι έχουμε ε, αυτή τη συμφωνία με το Πακιστάν θα είναι πολύ σημαντικό και για την ε, συνέχεια των συζητήσεων με την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας απεισδοχής, δεν θα σας εκπλήξει ότι είναι μια πολύ απλή συμφωνία. Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις επανεισδοχής για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τους υπηκόους της χώρας και τους απάτριδες έχετε τις συνήθεις διατάξεις σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διατάξεις για την επιστροφή των ανθρώπων στο Πακιστάν. Η εντολή είναι πολύ παλιά, όπως σας είπα στην αρχή, και είναι μια εντολή που δόθηκε με βάση το παλιό καθεστώς πρώτης Λισαβόνας είναι προφανώς, προφανές ότι όταν η Κομισιόν λάβει νέες εντολές από το Συμβούλιο ή όταν θα εξεταστούν οι νέες εντολές για τις συμφωνίες επανειδοχής, η Κομισιόν θα σεβαστεί πλήρως τους κανόνες που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόεδρε, όπως σωστά είπατε, το άρθρο 218 και η παράγραφος 10 όλες ιδιαίτερως αναφέρεται σε αυτά τα θέματα της εντολής. Αυτή είναι μια σύντομη παρουσίαση ε, ξέρω ότι λάβατε το κείμενο της Συμφωνίας Επανεισδοχής και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιασδήποτε ερωτήσει έχετε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο λόγος ε, στους εκπροσώπους της Προεδρίας. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπε η Κομισιόν. Όντως ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και γι' αυτό το λόγο στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν κάποιες τελευταίες διαφορές και δυσκολίες που είχαν απομείνει. Προβλέπεται εδώ πέρα μία αίτηση, ένα αίτημα διαβούλευσης και προβλέπεται επίση και μια διαδικασία σύμφωνη γνώμη συνένεση από το Κοινοβούλιο που έχει ξεκινήσει. Βάσει του άρθρου 119 τη συνθήκη για την Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Μπουζούτιλ, θέλετε εσεί το λόγο. Μπορείτε να μιλήσετε εξ ονόματο του κυρίου Σόγκορ. Ναι, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματο του κυρίου Σόγκορ, ο οποίο έπρεπε να φύγει, έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο, έχει μια πτήση. Δεν μπορούσε να παραμείνει λοιπόν τον αντικαθιστό να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπός ιδιαίτερα, ο οποίος ήρθε εδώ για να μας δώσει τις σημαντικές αυτές πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις. Σαφώς θεωρούμε ότι η συμφωνία επανεισδοχής με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με το Πακιστάν, είναι συμφωνίες πολύ σημαντικές Επομένως, ε, επί της ουσίας ε, είμαστε υπέρ των ε, αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων. Στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές. Επίσης, σημειώνω τα όσα είπε ο κύριος Μπός για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι σχετικές διατάξεις προβλέπονται συμφωνία καθιστούν συμφωνία πιο ενδιαφέρουσα και ουσιαστικά ενδυναμώνεται τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διαπραγματεύεται με άλλες τρίτες χώρες και συγκεκριμένα με την Τουρκία. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία που ακολουθείτε, από ό,τι κατάλαβα το Συμβούλιο δεν έχει, ε, μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει ακόμα την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου και το σημειώνω αυτό με ιδιαίτερη απογοήτευση. Όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι ε, και εμείς θα πρέπει να ενημερωνόμαστε όσο καλά ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο και την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Σεσίλια Μάλστρομ αυτό ακριβώς είπε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει την ίδια πληροφόρηση, την ίδια ενημέρωση, τα ίδια έγγραφα με αυτά που λαμβάνει το Συμβούλιο. Αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν έχουν να κάνουν συγκεκριμένε παρατηρήσεις, τότε θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Σόγκαρ μου ζήτησε να σας ενημερώσω ότι μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φως για την συμφωνία αυτή και μπορεί να αποσταλεί στην Ολομέλεια χωρίς να γίνει άλλη συζήτηση στην Επιτροπή μας. Από ό,τι φαίνεται όμως ακόμα θα πρέπει περιμένουμε την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Και κάτι ακόμα, ενδεχομένω αυτό να αποτελέσει ε, ερώτημα που θα μπορούσε να απαντήσει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως θα πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ίδια συμφωνία όσον αφορά το Κοινοβούλιο του Πακιστάν Ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα επικυρώσει συμφωνία αυτή το Πακιστάν, επομένως θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει και για αυτό το ζήτημα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Now. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να σχολιάσει. Ίσως καταρχάς ε, τα μέλη της Επιτροπής, εν συνεχεία Ξανά θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν και στην ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Κύριε Γκυγιόμ, λοιπόν, πρώτη από όλου. Κυρία Έντστα ή κυρία Γκυγιόμ. Κυρία Γκυγιόμ, ευχαριστώ. Δεν ήμουνα η πρώτη, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Ε, Όντω, καθυστερήσαμε. Τρία σχόλια θέλω να κάνω. Ε, Καταρχά, για το θέμα τη διαδικασία. Μα ε, ζητάτε να αποφανθούμε για αυτή την ε, συμφωνία. Υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2009, από ό,τι κατάλαβα. Στο μεταξύ, η συνθήκη της Λισαβόνας ε, τέθηκε σε ισχύ όπως υπενθυμί, μας υπενθύσατε. Ε, οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου σε μια προηγούμενη ε, συνεδρίαση μας είπαν ότι αυτές οι διεθνείς συμφωνίες που δεν εφαρμόζονται ακόμη θα πρέπει να εξεταστούν από το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της νέας διαδικασίας. Θα μπορούσαμε να μας διευκρινίσετε αυτό το πράγμα, θα μπορούσατε να μας πείτε τι ρόλο πρέπει να παίξουμε για αυτή τη συμφωνία. Τώρα, επί της ε, αρχής αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Έχω κάποια ερωτηματικά. Ε, στην πράξη, παρότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες ε, συμφωνίες, δεν εφαρμόζονται, εν περιπτώσει. περισσότερο οι διμερείς συμφωνίες εφαρμόζονται. Θα ήθελα να μου δώσετε λοιπόν, για να γίνει μια σωστή συζήτηση, κάποιες πληροφορίες για αυτά τα άτομα τα οποία εστάλησαν πίσω σε αυτές τις χώρες προέλευσης και διέλευσης ε, δυνάμει αυτών των συμφωνιών επανειστοχής. Ε, υπάρχουν ε, δυνατότητες ένταξης. Πώς μπορεί να γίνει. Ε, και τελευταίο στοιχείο για το Πακιστάν τώρα πιο συγκεκριμένα. Θα ξέρετε ότι είπα, η αρμοστία ε, παρενέβη πολύ περισσότερο τους τελευταίους μήνες γιατί υπήρξαν μετακινήσεις πληθυσμών αρκετά σημαντικές ε, λόγω των στρατιωτικών παρεμβάσεων στο Πακιστάν. Και με βάση τα στοιχεία που έχω, περίπου ένα εκατομμύριο άτομα έχουν εκτοπιστεί για τον ένα τον άλλο λόγο στο εσωτερικό αυτής της χώρας. Έχετε λάβει υπόψη αυτήν την κατάσταση ε, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας επανεισδοχής και αν ε, υπάρχουν ε, πολύ, σοβαρές, ε, πολύ σοβαροί λόγοι που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει απειλή για τη ζωή αυτών των ανθρώπων, υπάρχει περίπτωση να αναστείλουμε την εφαρμογή και την εκτέλεση αυτών των συμφωνιών. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω το εξής ερώτημα. Τις εξής ερωτήσεις φαίνεται να υπάρχει μια ανερχόμενη τάση για τους μετανάστες που έρχονται από το Πακιστάν. Έχει αυξηθεί βέβαια ο ρυθμός έλευσής τους και βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία μορφή ελέγχου της ε, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περίπτωση αυτών, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ανερχόμενη τάση έλευσης ε, μεταναστών από το Πακιστάν, οι οποίοι έχουν έρθει ως ε, πρόσφυγες ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Επίσης, ο Διεθνής Σύνδεσμος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει ζητήσει να μην υπάρξει συμφωνία με τον Πακιστάν στα θέματα αυτά, γιατί δεν υπάρχει, συμφω... δεν υπάρχει σεβασμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ποια είναι η θέση της ε, Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Και τέλος, σε σχέση με τον Πακιστάν και την προστασία των δεδομένων. Υπάρχει η πρόβλεψη να υπάρξουν μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να υπάρξει αυτή η προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Και πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ο αρμόδιος για την προστασία των ατομικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Vielen Dank. Signor Romeva. Madame Flotre. Madame Flotre. C'est compliqué aujourd'hui, hein, la parole. Περίπλοκο. Ποιο, το ποιο έχει το λόγο τελικά. Τα μπερδεύετε πολύ, Πρόεδρε, σήμερα. Α, νόμιζα ότι ήταν ο κύριο Τζομέβα. Ε, είναι πολύ ευγενή ε, ο κύριο ε, Ρωμέβα, γιατί πραγματικά έχει ζητήσει το λόγο. Μέχρι να πάω και να έρθω εγώ. Λοιπόν, η ε, Συμφωνία ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Πακιστάν. Είναι η πρώτη συμφωνία επί τη οποία μπορούμε να ασκήσουμε την κοινοβουλευτική μα αρμοδιότητα πλήρω, όχι πλήρω 100% και δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε. Αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένω να πούμε όχι και με βάση την αρμοδιότητά μα μπορούμε να ε, έχουμε παρέμβαση πριν υπογραφούν, δηλαδή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, πριν υπογραφούν οι συμφωνίε, αλλά και κατά τη διάρκεια τη εφαρμογή του γιατί στη μεικτή αυτή επιτροπή ε, για τις συμφωνίες αυτές δεν υπάρχει ρόλος για τους ε, βουλευτές. Αυτή είναι η Γενική Συμφωνία για τις Συμφωνίες Επανεισδοχής. Ε, αυτή η συμφωνία με το Πακιστάν είναι η πρώτη μετά τη θέση ισχύ τη Λισαβόνας. Αυτό που μας εκπλήσει είναι η πρώτη φράση της συμφωνίας. Η πρώτη φράση μιλάει για μια συμφωνία η οποία συστήνεται στο σχέδιο δράσης για το Αφγανιστάν που είχε παρουσιαστεί το 1999. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει συμφέρον για την Ευρώπη να ξαναστείλει στο Πακιστάν Αφγανούς οι οποίοι έχουν διέλθει μέσω του Πακιστάν. Έχουν διέλθει μέσω του Πακιστάν για να φτάσουν στην ε, Ευρώπη. Μετά περιπλέκονται ακόμα τα πράγματα. Γιατί αν κοιτάξετε, ποια άτομα αφορά αυτή η συμφωνία επανεισδοχής, ε, διερωτάστε μήπως απλώς θέλουμε να κάνουμε συμφωνίες επανειλικής μόνο και μόνο για να τις κάνουμε ε, ή έχουν πραγματική αποτελεσματικότητα οι συμφωνίες επανεισδοχής για αυτούς που τις θέλουν, γιατί εγώ δεν τις θέλω ούτως ή άλλως. Αν διαβάσετε καλά, βλέπετε ότι για να σταλεί το, το άτομο στο Πακιστάν δυνάμει αυτή τη συμφωνία επανεισδοχής, πρώτον, τα άτομα τα οποία είναι, πρέπει να είναι σε μη νόμιμη κατάσταση στο Πακιστάν και δεύτερον, τα άτομα τα οποία πέρασαν κατευθείαν από το Πακιστάν και ήρθαν απευθεία από το Πακιστάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, υπάρχει μια σχέση με την Τουρκία. Και είναι η σχέση με την Τουρκία. Ότι οι Αφγανοί περνάνε από χερσαίε οδού από την Τουρκία και όχι ε, με αεροπλάνα. Νομίζω ότι, ότι αυτή η συμφωνία θα ενταχθεί στο σχέδιο δράσης για το Αφγανιστάν. Αυτό μου φαίνεται περίεργο. Όταν βλέπουμε την συμφωνία ε, και την πραγματική τη σημασία, νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματική στρέβλωση ε, για αυτή τη συμφωνία. Κομισιόν, μπορείτε να μα πείτε ε, τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία. μα είπατε ότι συλλάβαμε 13.500 άτομα από το Πακιστάν με τι ε, προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία επανεισδοχή. Δηλαδή, φτάσανε απευθεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να φτάσουν καθόλου μέσω μια τρίτη χώρα. Ή όχι. Πρέπει να μα απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ποιον αφορά αυτή η συμφωνία επανεισδοχής, ποια άτομα αφορά και γιατί τη διαπραγματευθήκατε και γιατί θα εφαρμοστεί. Επίση, υπάρχουν ούτω ή άλλω προβλήματα με συμφωνίε επανεισδοχής εν γέννη. Ε, όποιον βουλευτή και να ρωτήσετε, δεν υπάρχει ένα που να μην σα πει μια ιστορία ε, που να έχει επαναπροωθηθεί σε μια χώρα δυνάμει μια συμφωνία επανεισδοχή και όπου εκεί, α πούμε, τον βασάνισαν, τον φυλάκισαν καταχρηστικά κτλ. Έχουμε ένα πρόβλημα δικαίου με τι συμφωνίε επανεισδοχή. Ε, λόγω τη αρχή τη μη επαναπρόθεση και τι διαδοχικέ ευθύνε που επισύρονται. Σε αυτή τη νέα εποχή κοινοβουλευτική ευθύνη που ανοίγει με τη Λισαβόνα, θα θέλαμε τώρα να ξεκινήσουμε από μια βάση αξιολόγηση σωστή και κοινή των συμφωνιών επανεισδοχή. Δηλαδή, οι ισχύουσε συμφωνίε επανεισδοχή μα οδήγησαν σε πόσα άτομα που τα στείλαμε πίσω και πώ σεβόμαστε την αρχή τη μη επαναπρόθεση. Εγώ δεν έχω ιδέα. Έχω ακούσει διάφορε προσωπικέ ιστορίε, αλλά δεν έχω έτσι μια στατιστική, μια σοβαρή ανάλυση. Αν κάποιο ξέρει, αν η Κομισιόν ξέρει, αν το Συμβούλιο ξέρει, αν υπάρχει μια μελέτη, με ενδιαφέρει τα μάρλα. πριν προχωρήσουμε, νομίζω θα πρέπει να μα πείτε πολύ συγκεκριμένα γιατί μιλάμε εδώ πέρα και τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή με αυτέ τι συμφωνίε επένδυση. Τι έχουμε πετύχει. Ζανίν Χένι Πλάσερ, θέλετε το λόγο. Και υπάρχει κανεί άλλο που θέλει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε και ο κυρία Φλότρα. Νομίζω ότι η Συμφωνία Επανεισδοχής είναι πάρα πολύ σημαντική και θέλουμε όντως να αρχίσει να ισχύει η Συμφωνία αυτή. Πέρασε πάρα πολύ καιρό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οι συμφωνίες αυτές είναι πολύ σημαντικές γιατί οι διμερείς συμφωνίες είναι αν θέλετε μία προσέγγιση βραχυπρόθεσμης επένδυσης, χωρίς όμως να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτά αποτελέσματα στο απότερο μέλλον. Ξέρετε βέβαια ότι σαφώς τίθενται κάποια νόμιμα ερωτήματα, σαφώς θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, πάντως εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας αυτής. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει το λόγο, τότε να δώσουμε πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στην Προεδρία και μετά στον Σάιμον. Πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τίθενται τρία ερωτήματα αυτή τη στιγμή, δύο γενικέ ερωτήσει. Η πρώτη έχει να κάνει με την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαπραγματεύεται τη συμφωνία αυτή και πώς θα εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να επαναλάβουμε μετά όσα είπαμε στην αρχή Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει και το Συμβούλιο. Η δεύτερη ερώτηση, να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ με τις απόλυτα δικαιολογημένες ερωτήσεις όσον αφορά την πολιτική επιστροφής ε, επαναπρόθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, όπως γνωρίζετε, ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει και να προχωρήσει σε κάποιες συστάσεις για τις πολιτικές αυτές. Επομένω, α μην υπάρξει καμία παρανόηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι ότι εκτελεί την εντολή που τη έχει δώσει το Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί μια συμφωνία επανεισδοχή με πολλέ χώρε, τρίτε χώρε αν είμαστε σοβαροί στην καταπολέμηση της ε, παράνομης μετανάστευσης και νομίζω το είπαν αυτό και οι υπουργοί που ήταν εδώ πέρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί λοιπόν στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη, τότε συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα της πολιτικής μας. Το τρίτο ερώτημα που ετέθη είναι αν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί ή όχι με την ε, Συμφωνία Επανεισδοχής ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Πακιστάν που είναι επιτάπητος αυτή τη στιγμή. Δύο λοιπόν γενικές ερωτήσεις και μία πιο συγκεκριμένη. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με την προτινόμενη Συμφωνία Επανεισδοχή μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και του Πακιστάν. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί μπορούμε να απαντήσουμε σε όλε αυτέ τι ε, δικαιολογημένες γενικές ερωτήσεις. Θα χρειαστούμε δύο ώρες όμως για να σας δώσουμε απαντήσεις. Εσείς θα αποφασίσετε θα το κάνουμε αυτό ή όχι. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, τότε και χρειαστεί να έρθουμε εκ νέου σε επαφή με το Πακιστάν, τότε ενδεχομένως να μην έχουμε στο τέλος καθόλου καμία συμφωνία επανεισδοχής. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση του Πακιστάν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις απέναντι στην πακιστανική πλευρά. Αν πάμε τώρα πίσω στο Πακιστάν και τους πούμε κοιτάξτε πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις από την αρχή, τότε θέτουμε εν κινδύνο την ίδια τη συμφωνία επανεισδοχής. Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Εμεί μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση εφόσον το επιθυμείτε. Uh, να σα υπενθυμίσω. Η Κομισιόν πάντα μπορεί να υποβάλει γραπτός πολύ πιο συγκεκριμένες ε, απαντήσεις ε, ή σχόλια σε κάθε μία από τις ερωτήσεις που έχουν ε, διατυπωθεί. σε όλες τις ερωτήσεις που έκαναν οι βουλευτές, αν δεν έχουμε τώρα τον απαραίτητο χρόνο να, το συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα εδώ, θα μπορούσατε κάλλιστα να απαντήσετε γραπτός, με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε, ακόμη και με εμπιστευτικό. Να δώσετε όλα τα στοιχεία που σας ζήτησαν οι βουλευτές. Γιατί αυτά τα στοιχεία χρήζουν προσοχής από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Εδώ βλέπω σηκώμενα χέρια. Αν δεν θέλετε να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση τώρα, σας κάνω έκκληση να είστε πολύ συνοπτικοί. Κυρία Φλότχα, ε, πολύ σύντομη. Ε, απαράδεκτη απάντηση. Έχω σκανδαλιστεί. Η Κομισιό λέει, ε, μπορώ να απαντήσω, αλλά δεν απαντάτε. Ε, απαντήστε λοιπόν, σας παρακαλούμε. Και αφήστε, σταματήστε αυτούς τους εκβιασμούς. Εάν δεν δεχθείτε αυτή την συμφωνία πάρα αυτά, ας πούμε, ε, ακυρώνεται. Αυτό είναι η συζήτηση. Αυτή είναι απαράδεκτη απάντηση. Merci. Ευχαριστώ. Κύριε Άνστ. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Χωρίς μικρόφωνο. Μακριά και χωρίς το μικρόφωνο. Θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε η κυρία Φλότρο. Η μόνη απάντηση η οποία δόθηκε είναι ότι υπάρχουν προβλήματα με το Πακιστάν. Φυσικά υπάρχουν μεγάλε ανησυχίε από διεθνεί φορεί, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει καταδίωξη για θρησκευτικού λόγου, για λόγου σεξουαλική ε, κατεύθυνση και για άλλου λόγου. Και δεν μπορούμε εμείς απλώς να πούμε ότι α, δεν έχουν καμιά σημασία όλα αυτά. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε επί αυτής της ε, βάσης. Αυτή η συμφωνία είναι πια ξεπερασμένη τη στιγμή που έχουν ανακύψει τόσο σοβαρά ερωτήματα. Ευχαριστώ. Η Καρίν, επειδή τρέχει ο χρόνος, και επειδή τα ερωτήματα αυτά πρέπει να τύχουν απαντήσεων, μήπω μπορεί η Κομισιόν να μα δώσει γραπτέ απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Και πάλι, εγώ δεν είμαι εδώ για να υποστηρίξω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εργάζεται επί του θέματο αυτού για χρόνια. Εμένα μου εξηγήσανε λεπτομέρειε και του, τους λόγους για αυτά τα θέματα σε ό,τι αφορά το Πακιστάν. Ίσως μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια διμερή επαφή με την Κομισιόν Ίσως η Κομισιόν να μας απαντήσει εγγράφος και προβούμε σε αυτές τις επαφές. Θα επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σταθώ σε δύο γενικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ερωτήσεων που διατυπώθηκαν. Δεν έχουμε τώρα τις στατιστικές που ζητούν τα αξιότιμα μέλη, αλλά Καταρχήν το θέμα της χρησιμότητας των συμφωνιών επανειστοχής. Βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο εφαρμογής αυτών των ε, συμφωνιών. Λίγα χρόνια μονάχα λειτουργούν αυτές οι συμφωνίες. Έχουν θετικό χαρακτήρα γιατί επιλύουν τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και οι επερχόμενες συμφωνίες οι οποίες θα εγκριθούν βελτιώνονται κάθε φορά σε κάθε βήμα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από την Κομισιόν και το Συμβούλιο από κοινού για να πετύχουμε αυτό το στόχο να αναβαθμίσουμε το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών. Επιτρέψτε μου να είμαι αισιόδοξο σε σχέση με την χρησιμότητα αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής. Εξάλλου θα ήθελα να σας ζητήσω να μην θεωρηθούν αυτές οι συμφωνίες επανεισδοχής σαν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο είναι στην πραγματικότητα. Είναι απλώς ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει να ληφθεί η απόφαση επιστροφής των μεταναστών που έχει ήδη ληφθεί βάσει των διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών σε κάθε χώρα. Αυτό σε ό,τι αφορά αυτό που αφορά τώρα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θέματα προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων, δεν νομίζω ότι στη διαδικασία επανεισδοχής που πρέπει να ληφθούν αυτά υπόψη, αλλά στο προηγούμενο στάδιο που είναι η λήψη αποφάσεως για την επιστροφή των μεταναστών, υπάρχει εκεί η οδηγία για την, ε, για την επαν, επαν, επαναφορά των μεταναστών, έχουμε το κεκτημένο μας για το άσυλο, επομένως η διαδικασία επανεισδοχής δεν επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται για να επιστραφεί ή να μην επιστροφεί ένας μετανάστης σε τη χώρα προέλευσή του. Σίμων, θέλεις να κλείσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Κομισιόν, αλλά και τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την ε, σύντομη αλλά πολύ ζωντανή συζήτηση. Φυσικά καταγράφω κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν από κάποιους συναδέλφους. Επίσης καταγράφω ότι κάποιοι συνάδελφοι ε, μοιάζουν να είναι κατά των, της ιδέας των συμφωνιών επανεισδοχής επί της αρχής. Θα συμφωνήσω όμως με την Ζανίν Χάνης Πλάσχαρτα με όλες τις παρατηρήσεις <coughs> και συμφωνώ ότι είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία αυτή που έχουμε μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ε, αν κατάλαβα καλά, εξορισμού, όταν μιλάμε για μια συμφωνία επανειστοχής, μιλάμε για υπηκόστη των χωρών που διαμένουν παρανόμως και που έχουν ήδη περάσει από τη διαδικασία ασύλου, ε, έχει απορριφθεί η αίτησή τους και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παραμείνουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επικράτειά της και επομένως η αρχή τη μη επαναπρόθεση δεν υπησέρχεται καθόλου εδώ. Το συντομότερο λοιπόν ε, περάσει αυτή η συμφωνία και αρχίσει να εφαρμόζεται τόσο το καλύτερο. Εκ μέρου τη Επιτροπής ε, θυμίζω τη σημασία της γραπτής απάντησης στα διάφορα σημεία και διάφορε ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί προς την Κομισιόν ή προς άλλους που δεν έχει, δεν έχει μπορέσει λόγω έλλειψη χρόνου η Κομισιόν να απαντήσει. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μα δίνετε ξανά το λόγο. Να μην μα παρεξηγήσετε, σα παρακαλώ. Εμεί θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σοβαρή και με κάθε σοβαρότητα ερχόμαστε εδώ. Έχουμε ακούσει πολλέ ερωτήσει που πραγματικά πρέπει να συζητηθούν σοβαρά μεταξύ τη Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είμαστε έτοιμοι για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι επίση να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να έχετε γραπτό και προτείνω επίση να γίνει μια συνάντηση μεταξύ της Κομισιόν και των εμπειρογνωμόνων της και του εισηγητή, ούτω ώστε όλες οι ερωτήσεις, ακόμα και αυτές τη κυρία Φλότχο και άλλων συναδελφών και άλλων βουλευτών, να απαντηθούν, αλλά μέσα σε κάποια χρονικά πλαίσια λογικά. Γιατί είναι περίπλοκα. Δεν είναι ότι δεν σεβόμαστε το Κοινοβούλιο, δεν πρόκειται περί αυτού. Ε, είναι ουσιαστική αυτή η συζήτηση για και τα ερωτήματα που, που θέσατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος, το καταγράφουμε. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο προς το παρόν και πάμε στο επόμενο σημείο. Μην ξεχνάμε και την συνέντευξη των συντονιστών αμέσως μετά. Το επόμενο σημείο είναι το σημείο 5, λέει ο Πρόεδρος, συμμετοχή της Ελβετίας και του Λίχτενστάιν στις ε, δραστηριότητες του Frontex. Uh, Θα ξέρετε ότι για αυτή τη συμφωνία υπάρχει μια διαπραγμάτευση εν εξελίξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελβετίας και του Λίχτενστάιν για τη συμμετοχή των διεθνών χωρών στις δραστηριότητες της Frontex. Η Κομισιόν θα, θα πάρει τον λόγο καταρχήν, εν συνεχεία η Προεδρία του Συμβουλίου και τέλος ο εισηγητής, ο κύριος Κλάης. Ε, η κυρία Μόνικα Μοσχάμερ, εκ μέρους Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με διαδικαστικά ζητήματα. Να αναφερθώ στην ημερομηνία απογραφή τη συμφωνία 30 Σεπτεμβρίου υπεγράφει, δηλαδή πρωτού αρχίσει να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα και η απόφαση ε, σύναψης της ε, συμφωνίας αυτής ε, ετέθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της διαβούλευσης μόνο. Θα αλλάξει όμως τη διαδικασία με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσετε την έγκρισή σας. Μέχρι στιγμής οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο προσπαθούν να προσαρμόσουν την συμφωνία αυτή προκειμένου να συνάδει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Προφανώς όμως θα ζητηθεί η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επί της ουσίας τώρα, η Ελβετία και το Λίχτενστάιν είναι τρίτες ε, χώρες συνδεμένες με τη Συμφωνία Σέγγεν και ως εκ τούτου υποχρεούνται να εφαρμόσουν όλες τις διατάξεις του κεκτημένου Σέγγεν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχουν και οι δραστηριότητε Frontex. Για ποιο λόγο όμω χρειαζόμαστε ξεχωριστή συμφωνία. Χρειαζόμαστε ξεχωριστή συμφωνία γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία του κανονισμού Frontex που δεσμεύουν τα δικά μας κράτη-μέλη μέσω του παράγου δικαίου και κατά αυτόν τον τρόπο δεν δεσμευόντουσαν χώρες όπως η Ελβετία και το Λιχτενστάν. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να υπογραφεί μία νέα συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 21 του καονισμού Frontex. Ήδη χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα στο παρελθόν με την Ισλανδία όταν υπογράψαμε μαζί τη συμφωνία το 2007. Τίποτα το νέο λοιπόν όσον αφορά την συμφωνία αυτή με την Ελβετία και το Λίχτενστάιν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε ακριβώ την ίδια γραμμή που είχε ακολουθήσει και στο παρελθόν. Προβλέπονται νέες διατάξεις για τα δικαιώματα ψηφοφορίας που μπορούν να έχουν οι χώρες αυτές στα πλαίσια του Frontex, προβλέπονται όμως και διατάξεις για, για το προσωπικό, καθώς επίσης και για την χρηματοδότηση που θα προέλθει από τις χώρες αυτές. Και τέλος να σας πω ότι το Liechtenstein συμμετέχει ήδη μολονότι το πρωτόκολλο σύνδεσης για το Liechtenstein δεν έχει επικυρωθεί δεν θέλαμε, θέλαμε εδώ πέρα να αποφύγουμε να γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσει. Καταλαβαίνετε όμως ότι το Λίχτενστάιν θα καταφέρει να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Frontex από τη στιγμή που η βασική συμφωνία θα έχει υπογραφεί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εκ μέρους της Προεδρίας τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και για το προηγούμενο σημείο θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας για τις διαδικαστικές προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν για το ζήτημα αυτό μετά από την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας και απλώς ήθελα να τονίσω και πάλι την αναγκαιότητα να υπάρξει αυτή η συμφωνία για να μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων για τις χώρες που συμμετέχουν στο Σέγγεν στην περίπτωση της Frontex χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Κύριε Κλέης, ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ε, εκπρόσωπο της ε, Προεδρίας από το Συμβούλιο. Αυτά πάντα πολύ σημαντικά. Όσον αφορά τη διαδικασία, το νέο στοιχείο είναι ότι ε, εμείς συναποφασίζουμε πλέον εφόσον ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε σε όλα εκείνα τα σημεία που εξηγούν για ποιο λόγο υπάρχει εδώ πέρα μία περιορισμένη προσέγγιση. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως έγινε και με την Νορβηγία και την Ισλανδία, ακολουθούμε αντίστοιχη διαδικασία εδώ πέρα με την Ελβετία και το Λίχτενστάιν. δύο χώρες που ανήκουν, θα ανήκουν στη ζώνη Σέγγεν χωρίς να είναι κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή που θα ανήκουν στο χώρο Σέγγεν θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρω το κεκτημένο Σέγγεν. Επομένως, είναι πολύ λογικό πιστεύω να πρέπει να συμμετέχουν τα κράτη αυτά και στις δραστηριότητε του Frontex. και να μπορούν δηλαδή να συνεργάζονται στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσουμε τη συνένεσή μας, τη σύμφωνή μας γνώμη για τη συμφωνία αυτή. Any Παρατηρήσεις υπάρχουν από άλλους, κύριε Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι και εγώ σύντομος. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τη συμφωνία αυτή και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία και ότι θα στηρίξουμε εμεί ω ε, Επιτροπή τη συμφωνία αυτή. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι ε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε τοπίσει κάποια προβλήματα με τη συμφωνία. Μία διευκρίνηση όμως θα ήθελα να μου δώσει ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ε, διαπραγματεύσεις με το Λίχτενστάιν για τη συμφωνία αυτή έχουν ολοκληρωθεί. Ας μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, γενικά σας λέω ότι είμαστε υπέρ της συμφωνίας αυτής. Και αυτό γιατί και βέβαια η Ελβετία και το Λίχτενστάιν βρίσκονται πολύ κοντά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι βέβαια και μέλη της ζώνης Σέγγεν. Επομένω, εμείς, τουλάχιστον η πολιτική ομάδα, είναι σαφώς υπέρ αυτής της συμφωνίας. Ο κύριος Κίρκ Χοπ. Κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να προσθέσω ότι εγώ είχα αναλάβει μια σειρά από εκθέσεις που είχαν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Ελβετία και το ακριτικό Λιχτενστάιν στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Με ενδιαφέρεται ιδιαίτερα αυτή η σειρά εξελίξεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ιδίω η Σουηδία θέλει να προχωρήσει περισσότερο στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμφιλεγόμενο μπορεί να είναι αυτό το θέμα σε ορισμένους ελβετικούς κύκλους, αλλά έχουν προχωρήσει στο Σέγγεν, έχουν προχωρήσει τώρα στο Frontex. Θα πρέπει να χαιρετήσουμε αυτή την εξέλιξη, σίγουρα η πολιτική ομάδα το πράττει αυτό, ενδιαμέσως όμως θα πρέπει να βοηθήσουμε ως δυνατόν περισσότερο την Ελβετία και το μικρό Λίχτενστάιν σε σχέση με άλλες δυσκολίες τους που συνάπτονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. να τους βοηθήσουμε λοιπόν και να τους παρατηρήσουμε να προχωρήσουν και περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις. Όχι. Τότε. Αν θέλει να πει κάτι η Κομισιόν, η Προεδρία, η Κομισιόν, κυρία Μάσχαμερ. Ναι, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να απαντήσω στον κύριο Μπούσουτιλ στο ερώτημά του οι διαπραγματεύσει με το Λίχτενστάιν για την Frontex έχουν περατωθεί, αλλά η συμφωνία πρέπει, δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή παρά μόνο όταν <clears throat> κυρωθεί το πρωτόκολλο συμμετοχής του Λίχτενστάιν στο Σέγγεν από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα δείτε λοιπόν και τις αποφάσεις αυτές, γιατί πριν από την, ε, ε, την εφαρμογή της συνδίκης δεν μπορέσαμε να κυρώσουμε την το μητρικό πρωτόκολλο για το Λιχτενστάιν ούτω ή Αλλά στι επόμενε εβδομάδε νομίζω θα γίνει αυτό πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Έχει να πει κάτι η Πρόεδρε? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Ωραία. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη διαδικασία. Περιμένουμε να μας δώσει η Κομισιόν νέα για τις εξέλιξεις. Κλείνουμε τη συζήτηση για τώρα και προσκαλώ τους συντονιστές να μείνουν στην αίθουσα στην συνάντηση των ιδίων αυτών συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ.